Καλημέρα σας στα ισπανικά και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Καθίστε σας παρακαλώ, γιατί θα αρχίσει η συνεδρίαση. Και έχουμε πάρα πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη, αμέσως μετά το καλοκαίρι. Καταρχάς ελπίζω να περάσατε καλά το καλοκαίρι όλοι σας. Να ξεκουραστήκατε να χαλαρώσατε και να φορτίσατε τις μπαταρίες σας και να είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ένα κτίριο λάκτισμα, πολύ βαριά συνεδρίαση, πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Σήμερα και αύριο έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα ακούσουμε την παρουσίαση της Φιλανδικής Προεδρίας. Θα ακούσουμε τους οργανισμούς που έχουν σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ακόμα και ψηφοφορία θα έχουμε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Παρακαλώ λοιπόν να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας αύριο πρωί-πρωί στις 9. Πουρνό, πουρνό. Έχουμε και κεκλεισμένο το θυρών μετά την τακτική συνεδρίαση την πρωινή σήμερα και συνεδρίαση των συντονιστών αργότερα. Αλλά ας αρχίσουμε ε, ως ήθιστε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, την οποία και έχετε στα χέρια σας για μπροστά υποθέτω. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές σχετικά με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ε, το πρώτο είναι έγκριση της ημερήσιας διάταξης, ωραία. Έχει ε, προσθεθεί ένα θέμα υπαριθμών 20. Μάλλον υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών. Είναι το PNR αυτό, αναβλήθηκε. Αν δεν διαφωνείτε, εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. the linguistic profile of this Έχουμε και ανακοινώσεις για το γλωσσικό. Έχουμε όλες τις γλώσσες σήμερα, εκτός από ε, λετονικά, γοεδελικά και μαλτεζικά. Συγγνώμη, ε, είναι γνωστό αυτό για όλη τη συνεδρίαση θα ισχύσει αυτό το γλωσσικό καθεστώς. Έχουμε και φιλανδικά το πρωί, αλλά όχι στις υπόλοιπες ε, συνεδριάσεις. Ωραία εγκρίνεται. Εγκρίνονται και ε, οι συστάσεις και αποφάσεις των συντονιστών βάσει του άρθρου 214 ε, του κανονισμού. Έχουμε μακρύ κατάλογο ορισμού εισηγητών, αλλά για να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω την παρουσίαση της Φιλανδικής Προεδρίας που έχουμε για σήμερα το πρώτο μας θέμα, Ξέρετε ότι κάθε 6 αλλάζει η προεδρία στο Συμβούλιο έχετε ένα κατάλογο ε, μακρύ ε, ε, συγγνώμη, εισηγητών που ενέκριναν οι συντονιστές και θεωρούμε ότι εγκρίνεται αυτός ο κατάλογος εάν συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ. Και πριν αρχίσουμε, επιτρέπω στον εαυτό μου, παίρνω το θάρρος, να σας επισήσω την προσοχή στην στο θάνατο του Τζάνι Μποταρέλη που ήταν ο επόπτης ε, προστασίας των πολιτικών δεδομένων. Λυπούμαστε πάρα πολύ που το χάσαμε. Εν ενεργεία ήταν. Επανειλημμένα τον είχαμε εδώ στη συνεδρίαση. Τον θυμόμαστε όλοι που μας ανέφερε για θέματα προστασίας δεδομένων που είναι τόσο προσφελή για μας και είναι... Ε, μάθαμε λοιπόν το καλοκαίρι ότι απεβίωσε Ε, έπασχε από βαριά ασθένεια και θα ήθελα να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στον ίδιο. Έχουμε και θέμα σήμερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα έρθει ο αναπληρωτή του, αλλά νομίζω καλό θα ήταν να ε, τηρήσουμε ενό λεπτού υγιής στη μνήμη του. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα διαβιβάσουμε τα συλληπιτήρια της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ στην οικογένειά του, όπως άλλωστε πράξαμε προσωπικά πολλοί από εμά και στον ίδιο το οργανισμό όπου υπηρέτησε, τον υπόπτη προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε και πάμε στο πρώτο θέμα για το επόμενο διάστημα δύο ώρες έχουμε παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Ε, θα λάβουν το λόγο οι κυρίες Άννα Μάγια Χέριξον, Υπουργός Δικαιοσύνης και Μαρία Οχαλό, Υπουργός Εσωτερικών. Σας θυμίζω ότι θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων για το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας από πλευράς των πολιτικών ομάδων. Είναι το τρέχον εξάμεινο βέβαια η Φιλανδική Προεδρία. Ε, οι συντονιστές λοιπόν θα πάρουν το λόγο σε μια πρώτη φάση για δύο λεπτά ο καθένας για να κάνουν ερωτήσεις και θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε και λίγο χώρο και χρόνο για τα υπόλοιπα μέλη, το πολύ 1,5 λεπτό, έτσι ώστε να προλάβουμε μέσα στο δύο ώρο που έχουμε προγραμματίσει. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης το χρόνο Πάντα πιέζει ο χρόνος. Έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε και όλους τους αρμοδίους για τους διαφόρους οργανισμούς που άπτονται το δικό μας θεμάτων. Όλοι θα έρθουν. Ο πρόεδρος, κάθε φορά εκτελεστικός διευθυντής, ποιο είναι το σχήμα του κάθε οργανισμού. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σήμερα και αύριο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το χρόνο. Θα ήθελα θερμά λοιπόν να καλωσορίσω και τις δύο κυρίες, και την κυρία Χένριξον και την κυρία Οχάλο. Θα ακούσουμε πρώτα τις παρουσιάσεις τους. 15 λεπτά, εκάστη. Το πρώτο ημίωρο θα είναι η δική τους παρουσίαση και μετά θα γίνουν ερωτήσεις από τους συντονιστές στον πρώτο γύρο. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πολιτικών ελευθεριών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Έχουμε μεγάλες προσδοκίε από την Φιλανδική Προεδρία και δεν είναι η πρώτη φορά που προεδρεύει η Φιλανδία και έχουμε εξαιρετικές αναμνήσεις ε, και εξαιρετική ανάμνηση από τον Ιούλιο που είχαμε ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών στο Ελσίνκι, εξαιρετική διοργάνωση, εξαιρετική φιλοξενία. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να ανταλλάξετε απόψεις με τα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, κυρία Χέριξον, Υπουργός Δικαιοσύνης, έχετε το λόγο. Very, Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, Λόπες Ακυλάρ, μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας σήμερα και είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες στα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων της Εφηλονδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέματα που έχουν ε, μεγάλη προτεραιότητα για εμάς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Και η μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες έδωσε σε εμά μια ισχυρή εντολή για τα επόμενα χρόνια, για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Η μεγάλη προσέλευση των πολιτών στις κάλπες είναι πάρα πολύ σημαντική για την δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ όλους εσάς για την ε, επιτυχημένη παρότρινση των πολιτών να ψηφίσουν. Το σύνθημα της Προεδρίας μας είναι «Βιώσιμη Ευρώπη, βιώσιμο μέλλον». Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να δώσει αποτελέσματα, αλλά μπορεί να το κάνει αυτό μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση αξιών. Η πρώτη προτεραιότητα της ε, Προεδρίας της Φιλανδίας θα είναι η δέσμευσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τις κοινέ ευρωπαϊκές μας αξίες. Το κράτος δικαίου είναι εκείνο που κρατά την Ευρώπη ενωμένη και επηρεάζει κάθε πτυχή της από τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εύρυθμη ενιαία αγορά. Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών και των επιχειρήσεων και αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα της Ευρώπης. Για τους λόγους αυτούς η Φιλανδία θέλει να ενισχύσει την εργαλειοθήκη για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Φιλανδία λοιπόν ε, καλωσορίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την δημιουργία ενός ε, ετήσιου μηχανισμού αναφοράς με στόχο την επίτευξη των ε, στόχων που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχουν συνεισφέρει πολύ σημαντικά στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρεί το κράτος δικαίου. Με τις εκθέσεις και τα ψηφίσματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έσπρωξε έτσι ώστε να ψηφίσουμε μία πιο αποτελεσματική εργαλειοθήκη για το κράτος δικαίου. Και δεδομένου τούτου αποφασίσαμε η αρχή του κράτους δικαίου να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της ε, Συνόδου των Υπουργών Δικαιοσύνης τον Ιούλιο η αποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία και ποιότητα των ε, συστημάτων δικαιοσύνης είναι πολύ βασικές πτυχές ε, του κράτους δικαίου. Και η εφαρμογή όλων αυτών των αρχών θα έχει και αντίκτυπο στην γενικότερη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Φιλανδία λοιπόν είναι πεπισμένη ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ βασική για την εργαλειοθήκη του κράτους δικαίου. Η Φιλανδική Προεδρία επομένως θα εισέλθει σε διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της ε, χρηματοδότησης και του κράτους δικαίου. Το Ταμείο λοιπόν για τις ε, αξίες τη Ένωση θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο που θα στηρίξει τις οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών και θα προωθεί το κράτος δικαίου στους Ευρωπαίους πολίτες. Το άρθρο 7 ανήκει στην εργαλειοθήκη μας και έχει ενεργοποιηθεί διότι ήταν αναγκαίο. Η Φιλανδία λοιπόν θα συνεχίσει τις ε, διαδικασίες αυτές και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, με την Προεδρία του Υπουργού του Πουάινεν θα εποπτεύει συνεχώς την ε, κατάσταση με την Πολωνία και θα διεξάγει μια πρώτη ακρόαση με την Ουγγαρία το Σεπτέμβριο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι συνειφασμένα μεταξύ τους. και σύντομα θα κλείσουν 10 χρόνια από τότε που έγινε νομικά δεσμευτική η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι μία πολύ σημαντική έκφραση των ευρωπαϊκών κοινών μας αξιών και χρειάζεται να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους. Επίσης πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για περισσότερες ίσες ευκαιρίες και για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω τη δέσμευση της επόμενης Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει νομοθεσία που θα καταπολεμήσει τις διακρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρώνει το δρόμο έτσι ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα σε θέματα ισότητας και μη διακρίσεων. Η διαφθορά είναι επίσης κάτι που υπονομεύει το κράτος δικαίου. Η διαφθορά είναι κάτι που παραμένει πρόκληση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι που επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη. Αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και καθυστερεί την οικονομική ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς, επιθυμούμε το Συμβούλιο να διεξάγει μία επί της συζήτηση έτσι ώστε να ενταθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Κυρίες και κύριοι, οι κοινέ μας αξίες είναι μια αναγκαία βάση και για τις προσπάθειες που καταβάλουμε στον χώρο της ασφάλειας. Γι' αυτό χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Και αυτό είναι άλλη μια προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας την οποία ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Η εσωτερική ασφάλεια είναι ένα προϊόν μιας αλυσίδας ε, πράξεων, μιας αληθές δράσεων και φορέων η οποία πρέπει να είναι άρρηκτη. Διαφορετικά, οι προσπάθειές μας να καταπολεμήσουμε το διασυνοριακό έγκλημα όπως για παράδειγμα την ε, διακίνηση ανθρώπων, θα αποτύχουν. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αποτυχία. Χρειάζεται να επιτύχουμε και να σταματήσουμε τη διακίνηση ανθρώπων. Η δικαστική συνεργασία επίσης ε, μεταξύ κρατών μελών είναι επίσης αναγκαία, διότι για την ασφάλεια χρειάζεται μία αλυσίδα συνεργασίας στις ε, ποινικέ διαδικασίες. Χρειάζεται λοιπόν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θεωρείται ως ένα αναπόσπαστο βασικό κομμάτι της ώστε να διοριστεί ο Ευρωπαίος εισαγγελέα αυτό το φθινόπωρο κατόπιν συνένεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή γρήγορα. Η πρόληψη τώρα του εγκλήματος θα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας. Όμως, όταν τελείται μια αξιόπινη πράξη, θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας τραμμένη και στα θύματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, ως ε, Φιλανδική Προεδρία να συζητήσω με τους συναδέλφους μου, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, στηρίξουμε περισσότερο τα θύματα. Η Φιλανδική Προεδρία θα συνεχίσει επίσης τις εργασίες έτσι ώστε να δρομολογήσει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να δώσει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη Σύμβαση να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά τις ε, νομοθετικές εκκρεμότητες, το Συμβούλιο ήδη έχει υιοθετήσει μία θέση για την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ηλεκτρονική εγκληματικότητα και τώρα αναμένουμε την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η ψηφιακή επανάσταση επίσης έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συντελείται μια, ένα έγκλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση, την ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων με σεβασμό στα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρωτοπόρος ε, ό,τι αφορά τις προσπάθειες ε, υπεράσπισης της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρώπης. Αυτό θα φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Η Προεδρία λοιπόν της Φιλανδίας θα προωθήσει την διαφάνεια σε όλα τα θέματα τα νομοθετικά θέματα του Συμβουλίου και σε όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Επίσης, θα δημοσιεύουμε πληροφορίες για όλες ε, τις υπουργικέ διασκέψεις ε, μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας, καθώς επίσης και για τις συναντήσεις με τις ομάδες πίεσης, με τα λόμπι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας και πέρα από αυτή. Και με τα χαρά θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Εμεί σα ευχαριστούμε, Υπουργέ Χέρισον, και για την προσήλωση που δείχνετε στα θέματα που τόσο πολύ μα ενδιαφέρουν. Η σειρά σας τώρα, Υπουργέ Εσωτερικών, κυρία Οχάλο, για ε, το επόμενο τέταρτο, παρακαλώ. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Αξιότιμε Πρόεδρε. Ήταν χαρά μας ευκαιρία που είχαμε να συναντηθούμε στο Ελσίνκι πριν από λίγους μήνες και σας ευχαριστώ γι' αυτό αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι τιμή μου σήμερα ευκαιρία που έχω να σας απευθύνω το λόγο για τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Οι προκλήσεις και τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια είναι πολυπληθή και δεν γνωρίζουν σύνορα. Έχουμε την κλιματική κρίση, ε, στρατιωτικές απειλές, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές και ε, τους ε, πόρους που φθήνουν. Επίσης, το δημογραφικό, η κινητικότητα των πληθυσμών, τα λοιμώδη νοσήματα, το οργανωμένο έγκλημα και διάφορες απειλές. Αλλάζει λοιπόν το περιβάλλον χρειάζεται μια συλλογική και συνολική ε, προσέγγιση ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, πάρα πολύ διαφορετικές απειλές και πολυπληθής. Η κοινωνική διάσταση της ασφάλειας, μεταξύ αυτών η ε, συμπερίληψη και η ένταξη όλων των μελών δυνατών στην κοινωνία, η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων ε, παίζουν ε, ρόλο ζωτικό στην πρόληψη πολλών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι εκ των όνων κάνευ για να πληρούνται αυτά τα κριτήρια ασφαλείας. Η Φιλανδική Προεδρία έχει αρχίσει μια συζήτηση για το μέλλον της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά στοιχεία κλειδιά αυτής της συζήτησης είναι η ε, ενίσχυση της συνεργασίας των διοκτικών αρχών οι οργανισμοί ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζουν επίσης πρωταγωνιστικό ε, ρόλο. Η συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία των διοκτικών αρχών βασίζεται και στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα νέα συστήματα και με την πληροφορική. Χρειάζεται λοιπόν διαλειτουργικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η κείμενη νομοθεσία θα εφαρμόζεται. Η Φιλανδική ε, Προεδρία τονίζει και υπογραμμίζει ότι στη δικαστική συνεργασία κάθε ε, κρίκος της αλυσίδας ε, έχει σημασία για την εσωτερική ασφάλεια. Λαμβάνονται μέτρα για τη σωστή εφαρμογή των νόμων και θα πρέπει πάντα αυτά να λαμβάνονται υπόψη στη μελλοντική ε, ενίσχυση της συνεργασίας. Οι ικανότητες αντιμετώπισης υβριδικών απειλών θα πρέπει να ενισχυθούν και σε επίπεδο ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Οι φορείς της εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να αυξήσουν την αφεκτικότητα της κοινωνίας και την αντίσταση απέναντι σε διάφορες απόπειρες και απειλές. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τρόπο διαρθρωμένο και συντονισμένο. Η συντονισμένη δράση επίσης της Ένωσης χρειάζεται για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας κρισίμων υποδομών. Παρόλο που οι μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν, η απειλή παραμένει έντονη η Φιλανδική Προεδρία θα φέρει προς συζήτηση τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να προλαμβάνουν ε, το βίο εξτρεμισμό και να καταπολεμούν την ε, τρομοκρατία κάθε είδους και ιδεολογίας. Το φαινόμενο των ξένων μαχητών και ο τζιχαντισμός ε, είναι βασικές τρομοκρατικές απειλές, αλλά όχι μόνες. Οι τρομοκρατικές ε, απειλές από τη βία η άκρα δεξιά είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να προσέχουμε και να λαμβάνουμε υπόψη. Η πρόληψη της βίαιης ρίζοσπαστικοποίησης και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρειάζονται αλληλοϊποστήριξη. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στη σωστή ανάλυση και των απειλών και στα σωστά δεδομένα η Φιλανδική Προεδρία θα εστιάσει στην ε, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτσων που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της ε, ακραίας και βίαιης ρίζοσπαστικοποίησης. Θα πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε για νέες απειλές. Επιπλέον θεωρούμε σημαντικό να μην ε, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση στο διαδίκτυο για τρομοκρατία και άλλες παρανομίες το παράνομο περιεχόμενο στο ίντερνετ έπαιξε μεγάλο ρόλο στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είμαστε ε, δεσμευμένοι ε, να παρακολουθήσουμε ε, τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Η νομοθεσία θα πρέπει να είναι σαφέστατη, έτσι ώστε όλοι οι φορείς να γνωρίζουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς επίσης και να μπορούν να δρουν σε επίγουσες καταστάσεις. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ε, τους παρόχους υπηρεσιών ε, ίντερνετ. Οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες δεν χρησιμοποιούν μόνο τα αεροπλάνα για να ταξιδεύουν, αλλά και άλλα μέσα μεταφοράς. Για να μπορούν να διώκονται αυτές οι αξιόπινες πράξεις, θα πρέπει να δούμε μήπως ε, ε, υπάρχει δυνατότητα συλλογής PNR, προσωπικών δεδομένων επιβατών και σε άλλα μέσα μεταφοράς, πλην των αεροσκαφών. και στο σιδηρόδρομο και στην ακτοπλοεία. Θα πρέπει να το εξετάσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διασυνοριακή ε, θα πρέπει να δούμε και τις αναδυόμενες απειλές, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν νέες τεχνολογίες και να είμαστε προδραστικοί, ε, να προλαμβάνουμε, να προετοιμαζόμαστε. Η κυβερνοασφάλεια είναι σημαντικό στοιχείο για να ενισχύσουμε το ρόλο ε, της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καταπολέμηση της κυβερνο τρομοκρατίας και των απειλών χρειάζονται γρήγορες λύσεις και ταχεία απόκριση ε, από τις διοκτικές αρχές και από τις αρχές ασφαλείας. Στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία αποθηκεύονται και δίνονται στην αστυνομία το συντομότερο επιταχύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει βέβαια πάντα να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των κρατών μελών και ε, να είναι δεδομένη και να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Τεχνική νοημοσύνη, αυτοματοποίηση, νέα στοιχεία που είναι στην καρδιά της ανάπτυξης εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημόσιες αρχές μας. Η εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος ε, σε αυτά και οι ιδιοκτικέ αρχές και αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να διαθέτουν προηγμένα εργαλεία και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να εξετάσουμε την νομοθεσία και την ανάπτυξη των πόρων για να μπορούν να χρησιμοποιούν οι διοκτικές αρχές τις νέες τεχνολογίες ε, για να εξασφαλίσουν την εσωτερική ασφάλεια, σεβόμενες πάντα τις ε, ε, ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την ανάλυση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του δημοσιογράφους που ε, δολοφονήθηκαν. Και γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, είναι απαραίτητο να γίνει μια δημόσια έρευνα στην ε, Μάλτα για τις δολοφονίες αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να παρέχει ασφάλεια στην έρευνα, διάσωση και αποβίβαση και επίσης καταμερισμό ευθυνών με δίκαιο τρόπο σε όλα τα κράτη, ε, από όλα τα κράτη-μέλη. Η Μάλτα, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία δεν θα πρέπει να μείνουν μόνες τους σε αυτήν την προσπάθεια ε, και θα πρέπει να δοθεί βάση στην δημιουργία ενός προσωρινού ε, συστήματος μετεγκατάστασης. Γι' αυτό ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας ε, για να γίνει αυτός ο προσωρινός μηχανισμός μόνιμος και τι θα γίνει μέχρι να αναθεωρηθεί το, η νομοθεσία για το άσυλο. Η δέσμη μέτρων που είχε υιοθετηθεί αποδείχθηκε μη αποτελεσματική. Από την άλλη βέβαια το Κοινοβούλιο ακόμα περιμένει το Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του για τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του κοινού συστήματος ασύλου. Εσείς λοιπόν ως Φιλανδική Προεδρία θα μπορέσετε να πιέσετε τα κρατημέλη έτσι ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία μέχρι το τέλος της θητείας σας για να μην βρεθούμε πάλι σε αυτή τη δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζήπελ, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τις ε, δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις τους. Αναφερθήκατε στον τομέα της ασφάλειας. Να πω καταρχά ότι δεν έχει νόημα να ψηφίζουμε νέου νόμου αν δεν ε, έχουμε τη δυνατότητα να τους ε, εφαρμόσουμε μου φαίνεται πως ε, λείπει η πολιτική βούληση ε, για να γίνει αυτό ή ίσως το δικαστικό σύστημα και οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν την ε, νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτό. Μετά αναφερθήκατε σε γενικότερες κοινωνικές πτυχέ που αφορούν την ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω όταν μιλάτε για εντάξει, Θεωρείτε πως αυτό είναι μια πρόκληση που αφορά μόνο τις τρίτες χώρες, μόνο όσους έρχονται από εκεί. Ε, νομίζω πως υπάρχουν προβλήματα ένταξης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ορισμένους πολίτες της. Ε, είναι αυτό κάτι που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, να πω πως χαίρομαι πολύ που τονίσατε ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να θεωρούνται ε, ένα αναπόσπαστο σύνολο, κομμάτι της, ε, να θεωρούνται σύνολο. Αναφερθήκατε και στο άρθρο 7. Θα ήθελα λοιπόν να μας ε, ενημερώσετε για τις τρέχουσες εξελίξεις με την Πολωνία και την Ουγγαρία και το άρθρο 7. Επίσης, ποια είναι η δική σας άποψη για το αν ορισμένα κράτη-μέλη, πάνω από δύο, δεν ακολουθούν τους κανόνες, δεν σέβονται τα δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Εσείς ποια άποψη έχετε, θεωρείτε πως θα πρέπει να γίνουν περικοπές, να, να κλείσει η στρόφιγγα, να να μην δοθούν άλλα χρήματα. Επίσης, τι άποψη έχετε για την διεύρυνση του PNR σε άλλα μέσα μεταφοράς πέραν του ε, αεροπλάνου και ποια είναι η βάση αυτών των συζητήσεων. Πού στηρίζεται δηλαδή αυτή η πρόταση για διεύρυνση του PNR σε άλλα μέσα μεταφορά, Έχετε κάποιε αποδείξει για το ότι αυτό ήταν αποτελεσματικό, για παράδειγμα, στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία ε, και την καταπολέμηση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας. Πού βασίζεται λοιπόν αυτή η πρόταση για διεύρυνση του συστήματος PNR. Επίσης, αναφερθήκατε στο 5G και στην πρόσβαση των ε, αρχών επιβολής του νόμου σε αυτό. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με αυτό, τι σημαίνει δηλαδή ότι οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν το 5G. Ταυτόχρονα να πω ότι διάβασα πρόσφατα πως η Πολωνία υπέγραψε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το 5G. Αυτό πώς θα επηρεάσει το έργο μας και τι ακριβώς αποφάσισε δηλαδή, τι υπέγραψε η Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για την ομάδα Renew, κυρία Ιντφέλντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τις ε, δύο Υπουργούς Καλωσορίζουμε την Φιλανδική Προεδρία και τη φιλοδοξία ε, καθώς και την φρέσκια ματιά που ε, έχετε για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το κράτος δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως και για την ομάδα Renew. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πολύ που η Φιλανδική Προεδρία έχει τονίσει τη σημασία του. Και έχει αναγνωρίσει επίσης ότι υπάρχουν διάφορα θέματα με το κράτος δικαίου, διόλου ευχάριστα. Ε, μπορεί τα εθνικά μας συστήματα να διαφέρουν, μπορεί να έχουμε διαφορετικές παραδόσεις, όμως οι αξίες μας είναι κοινέ. Οι εθνικές ιδιαιτερότητες ε, είναι κάτι υπαρκτό, όμως υπάρχουν κοινά πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και βλέπουμε πως δεν εφαρμόζονται εξίσου σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Και φυσικά τώρα βλέπουμε τις δύο χώρες ε, για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 7, την Ουγγαρία και την Πολωνία, έχουν εκφραστεί ανησυχίε και για άλλε χώρε, όπω ακούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτόν τον νέο μηχανισμό ε, υποβολή αναφορών. Με τον κύριο Τίμερμανς συζητήσαμε την πρόταση αυτή. Εμείς όμως θα θέλαμε να τη δούμε πιο ενισχυμένη. Θα θέλαμε ε, μία πρόταση όπω αυτή που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογή. Είχαμε συντάξει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία ω απάντηση στην πρόταση τη Επιτροπής. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο. Έχετε την πρόθεση να συζητήσετε για το ενδεχόμενο ενό κοινού μηχανισμού για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά για έναν μηχανισμό για κάθε θεσμικό όργανο. Έχετε λοιπόν την πρόθεση να συζητήσετε ένα κοινό μηχανισμό με κοινά πρότυπα. Η Φιλανδική Προεδρία έχει σκοπό να συζητήσει το άρθρο 7 στέλνοντα μια επίσημη πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι κάτι που το περιμένουμε πολλούς μήνες τώρα. Τέλος, άσυλο και μετανάστευση. Δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα. Το Συμβούλιο επιτέλους πρέπει να λάβει αποφάσεις για τη δέσμη μέτρων ε, που καθυστερεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν κάνει το καθήκον του. Δεν κάνει αυτό που πρέπει. Ρίχνει τους πολίτες με αυτήν την κολυσιαρχία. Νομίζω πως πρέπει να πιέσετε το Συμβούλιο και εμείς ίσως θα έπρεπε να το πιέσουμε, να παγώσουμε το προϋπολογισμό του μέχρι να αναλάβει ευθύνε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στρίκ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τις δύο υπουργούς με τη σειρά μου για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Να σας ευχηθώ καλή τύχη για την Προεδρία σας και να σας συγχαρώ για το πρόγραμμά της. Επίσης, ε, γιορτάζουμε την 20η επέτειο των ε, συμπερισμάτων του Τάμπερε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Τι έχετε να πείτε για τους στόχους της, του Τάμπερε και για το αν έχουν επιτευχθεί στα 20 χρόνια που πέρασαν. Η κυρία Χισάνο ήδη ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία σε θέματα εσωτερικής διάστασης της μετανάστευσης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα για το Άσυλο. Αλλά φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία με τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να αποτραπεί η μετανάστευση και να υπάρξει συνεργασία σχετικά με, τα, ε, ε, με Οι πολιτικές αυτές όμως έρχονται είναι αντίθετες στο κράτος ε, δικαίου και στα θεμελιώδει αξίες της Ένωσης και η Ένωση θα πρέπει να ηγείται ε, σε όλους τους ε, σχετικούς τομείς. Αν δείτε τι γίνεται στη Λιβύη, είναι ένα φρικτό παράδειγμα. Οι μετανάστες είναι θύματα βίας. Και όμως, παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει το λιμενικό της Λιβύης να στέλνει πίσω τους μετανάστες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι έχουν κολλήσει κάπου στο ενδιάμεσο χωρίς να έχουν καμία πρόσβαση σε, στη διαδικασία ασύλου, χωρίς να έχουν καμία προστασία. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί τη Φιλανδική Προεδρία. Επίσης, ίσως η ε, κυρία Υπουργός θα μπορούσε να μας πει πώς... Ε, θεωρεί ότι θα διασφαλιστεί αυτή η συνεργασία να πηγαίνει χέρι με χέρι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα σέβεται. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ζητήσει κάποια εκτίμηση αντικτύπου, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποια θα είναι οι επιπτώσεις στους πρόσφυγες και του μετανάστε. Επίση, ε, τι άποψη έχετε για αυτόν τον μόνιμο μηχανισμό επιτήρηση και ελέγχου. Επίση, α είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για αρνητικά κίνητρα, εννοούμε τις κυρώσεις για τις τρίτες χώρες. Και αυτό λοιπόν είναι καλό να το λέμε. Ε, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τους άλλους στόχους ε, μας ό,τι φορά τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και να μην μένουμε μόνο στο μεταναστευτικό. Τέλος, να πω πως ε, μας ε, χαροποιεί πάρα πολύ η πρόταση για, για ενίσχυση των ε, νομικών διάβλων, έτσι ώστε η μετανάστευση να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της δική σα προεδρία. Η νόμη μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ε, έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. Το παρακαλώ να το έχετε υπόψη οι συντονιστέ και να τηρείτε το δίλεπτο. Η ομάδα ID, ο κύριο Σταρντίνου εδώ κάθομαι. Ε, Υπουργή είχε άνοιξον και εγώ χίσαλο. Ευχαριστώ. Σας έχω χαιρετισμού από τη συνάδελφό μας στη Φιλανδία και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην ε, Προεδρία, όπως και στην Εστονική πριν από δύο χρόνια. Έχω δύο ερωτήσεις για τις διάφορες πολιτικές που αναφέρετε. Το πρώτο είναι το κράτος δικαίου. Φυσικά, όταν υπάρχουν κανόνες θα πρέπει όλοι να του στηρούν όλα τα κράτη-μέλη. Δεν χωρά καμιά αντιβολία. Αλλά ταυτόχρονα μήπω βλέπετε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην πολιτική μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πρόκειται για το σεβασμό του κανονισμού του Δουβλίνου. Συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να σεβόμαστε και όλοι είναι υπεύθυνοι για τα εξωτερικά σύνορα και για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Σήμερα όμως βλέπουμε οργανώσεις πολιτικούς, ακόμα και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο να υποστηρίζουν στις ε, ομιλίες τους την παραβίαση του κανονισμού του Δουμβλίνου. Δεν το βλέπετε αυτό. Από τη μια λέμε ότι έχουμε προβλήματα με το κράτος δικαίου και θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και από την άλλη πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγουν ότι είναι πολύ ε, εντάξει να παραβιάζεται ένας κανόνας που είναι ο κανονισμός του Δουβλίνου. Δεύτερον, ακούσαμε πολλά εδώ για τη νέα συμφωνία ή το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Οι περισσότερες χώρες που είχαν την Προεδρία τα τελευταία χρόνια μας έταζαν ότι θα βρίσκανε τη λύση. Δεν τη βρήκαν ακόμα. Αν αυξηθεί πάρα πολύ η πίεση, μήπως υπάρχει κίνδυνος από αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, ας πούμε. Δηλαδή να μην είναι αρμόδια πλέον τα κράτη-μέλη για τα εξωτερικά του σύνορα. Αυτό δεν συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ μεγάλο. Και υπάρχει κίνδυνος να μιμηθούν το Brexit άλλα κράτη-μέλη. Και μια που μιλούμε για το άρθρο 7, τι λέτε για την Ουγγαρία, έχει δαπανίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τα εξωτερικά σύνορα. Ήταν καλή ιδέα ή όχι να επενδύσει εκεί. Και υποστηρίζεται και την ίδια πολιτική ε, την Ελλάδα, ε, την Ιταλία και άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Προφανώς, ε, αγαπητοί Υπουργοί, ο κύριος Μάντισον και όχι η συνάδελφός μου, η κυρία Αρταντίνο, είναι που εκπροσωπούν την ομάδα του IDEA. Τώρα όμως, να ακούσουμε την ομάδα του ECR, Πορκατσίνη. Είναι το όνομά σα. Ε? ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του υπουργού για την ε, παρουσίαση του σήμερα το πρωί και να κάνω ένα γενικό σχόλιο από πλευρά μου, αν μου επιτρέπετε. Πρόσεξα ότι το θέμα της διαχείρισης ε, της μετανάστευσης είναι εκτός των τεσσάρων βασικών πυλώνων σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που έχει προτείνει η Φιλανδική Προεδρία. Αυτό μας ανησυχεί λοιπόν. Γιατί η διαχείριση της μετανάστευσης, αν θεωρούμε ότι είναι εκτός της αίθουσα αυτής και πλήττει παράλληλα τόσο πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που ανακύπτει έχει να κάνει με τον μηχανισμό προσωρινής μετεγκατάστασης. ο οποίος αναφέρεται στο πρόγραμμα. Και εδώ θα ήθελα να υπάρχει μια σαφέστερη διάκριση. Να μην ε, κάνουμε παιχνίδι με τις λέξεις. Να σας πω το εξή η μετεγκατάσταση πάντα θα πρέπει να είναι προσωρινή. Δεν υπάρχει πιο προσωρινή της προσωρινής. Αυτό που θα ήθελα να αποφύγουμε, ωστόσο, θα ήταν ένα παιχνίδι με τις λέξεις για να μπαίνει κόσμους στην Ευρώπη και να λένε ότι έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν κυβεύεται το ποιο έχει δικαίωμα διεθνού προστασία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η επιλογή του ποιο έχει και ποιο δεν έχει δικαίωμα διεθνού προστασία έχει να κάνει με την χώρα προέλευση, όχι με τη χώρα προορισμού. Γιατί αυτό θεωρώ ότι μα προκάλεσε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Μία άλλη πολύ απλή ερώτηση για το κράτο δικαίου. Όλοι μας συμφωνούμε ότι το κράτος δικαίου έχει να κάνει με την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής κτλ. Όλοι συμφωνούμε για τα γενικά. Το πρόβλημα όμως ανακύπτει όταν το κράτος δικαίου χρησιμοποιείται ως πολιτικό επιχείρημα. Ένα αντικίνητρο για όσους έχουν διαφορετική αντίληψη από τη δική μας. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την δημοκρατία. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνης τώρα από την ΚΟΥ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και η δική μας ε, ομάδα εύχεται ότι καλύτερο για τη Φιλανδική Προεδρία. Έχω δύο θέματα που με απασχολούν. Καταρχάς, το θέμα του κράτους δικαίου. Τα λόγια είναι όλα φανταστικά και όμορφα για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας κάνουν περήφανος και ούτω καθεξής. Αλλά το θέμα είναι ότι ε, τηρούμε αυτές τις αρχές. Ε, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία, σε, σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε προβλήματα. Και πιστεύω ότι σε κάθε χώρα δηλαδή που θα κοιτάξουμε θα βρούμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του κρατού δικαίου. Αυξάνονται αυτές οι περιστάσεις. Έχω να ρωτήσει λοιπόν το εξή για τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χέντριξον, για την ε, αξιολόγηση και την διατήρηση του κράτου δικαίου. Ποια εργαλεία λοιπόν πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν. Τι θα κάνουμε με τους μεγάλους παραβάτες του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας λοιπόν συγκεκριμένα τι μέτρα θα έχετε υπόψη σας. Δεύτερο θέμα, φυσικά η μετανάστευση και εδώ θα στραφώ προς την κυρία Βυσάλο. Μιλήσατε πολύ για θέματα εσωτερικής ασφάλειας τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όπω είναι και θα ήθελα να μου πείτε το εξή σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι καταστροφική, όπω το ξέρετε. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του και εμεί καθόμαστε και κοιτάμε. Και 14 άνθρωποι βγήκαν και είπαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού. Εδώ λοιπόν τη Φιλανδική Προεδρία θα σε ό,τι αφορά τη συμμαχία των προθήμων των, ε, για την διάσωση ανθρώπων στην, Ευρω... στην Μεσόγειο. Θα τους υποστηρίξετε σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που χάνουν α, ε, τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Και για το κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου το Κοινοβούλιο υπέβαλε σχετική πρόταση. Για όλα φυσικά κάναμε πρόταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και δύο χρόνια. Περιμένουμε να κάνετε διαπραγματεύσεις μαζί μας. Θα κάνετε κάποιο βήμα προς την πλευρά του Κοινοβουλίου για το κοινό σύστημα χορήγηση ασύλου, προκειμένου να βρούμε ε, μια διαπραγμάτευση και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τώρα είναι η σειρά των συντονιστών. Έξι λεπτά να προτείνω. Τελείωσαν οι συντονιστέ. Να δώσουμε έξι λεπτά στου υπουργού ε, για να απαντήσουν. Για να ακούσουμε και του υπόλοιπου βουλευτέ στη συνέχεια. Η Υπουργό Χέντριξον είναι η πρώτη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μιλήσω σου ειδικά. Άρα σας παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Πόσο χρόνο έχω. Έξι λεπτά η κάθε μία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις που μου θέσατε. Και συχνά αναφερθήκατε σε θέματα κράτους δικαίου και χαίρομαι που το κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να ενισχύσουμε από εκείνου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να ενισχύσουμε και το κράτος δικαίου. Ζητήσατε συγκεκριμένες απαντήσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις κοινέ μας αξίες. Το κράτος δικαίου αποτελεί προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το μέλλον και τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν ε, απαραίτητο να προασπιστούμε αυτές τις κοινέ αξίες που ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που επιτρέπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί. Η Φιλανδία που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να δράσει ενεργά, να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα εργαλεία για την διατήρηση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε πιο προφανείς και αποτελεσματικές λύσεις για την υποστήριξη του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν η Φιλανδία θέλει να προωθήσει έναν τακτικό διάλογο σε ό,τι αφορά τέτοια καθημερινά ζητήματα, προκειμένου να είναι πιο εύκολο να διακρίνουμε τις τάσεις όπως διαμορφώνονται. Η Φιλανδία λοιπόν θα ήθελε να διεξαγάγει μια συζήτηση για το πώς ε, εξελίχθηκαν τα θέματα κράτους δικαίου και πώς στηρίθηκε το κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια στα κράτη-μέλη. Η έκθεση η οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση θεωρώ ότι αποτελεί ένα ενδεδειγμένο μέσο για να γίνει ακριβώς ο διάλογος αυτός. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη μα σε ό,τι αφορά την διατήρηση και την εγγύηση του κράτου δικαίου. Και εδώ αυτό εντάσσεται και στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη σύνδεση τη στήριξη του κράτου δικαίου με τη συνέχιση τη χρηματοδότηση. Τα γνωρίζετε άλλωστε αυτά. Δεν πρόκειται για μηχανισμό επιβολή κυρώσεων. Θέλουμε απλά να εξασφαλίσουμε ότι δεν γίνονται καταχρήσει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη εξίσου. Και σε ό,τι αφορά κάποια παραδείγματα. Να τονίσω επίσης ότι έχουμε πολλά μέτρα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ποια είναι τα μέσα αυτά και τα μέτρα αυτά. Τώρα, να περάσω στην Πολωνία και στην Ουγγαρία και το άρθρο 7. Σκοπός μας θα πρέπει να είναι ο εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον θα θέλαμε να μην χρειάζονται καν τέτοιε διαδικασίες. Θα θέλαμε να μπορούμε να προλαμβάνουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατά της Πολωνίας και κατά της ε, Ουγγαρίας και θα συνεχιστούμε, θα συνεχιστούν οι διαδικασίες αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλαβαίνω ποια είναι η δική σας ε, οπτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Ο συνάδελφό μου, ο Υπουργό του Πυράνινα, ο οποίο ε, είναι αρμόδιο για τέτοια θέματα στο Συμβούλιο, έχει συμφωνήσει άλλωστε για να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Και μπορώ λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι με τον τρόπο αυτό θα ακούσουμε και την δική σας φωνή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε το θέμα της διαφθοράς. Πώς μπορούμε να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Εδώ χρειαζόμαστε την υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα πρέπει να βρούμε λύσει. Γιατί και αυτό το χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε περιπτώσεις παραβίασης του κράτους δικαίου. Τώρα, σε διαφορά τα θέματα των, του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί προφανώς σε μια δημοκρατία επιβάλλεται η ελεύθερη χρήση του τύπου, η ελευθερία έκφραση της άποψης του καθενός. Αυτό μάλιστα κατοχυρώνεται και στις συμβάσεις, στις συνθήκες. Και φυσικά θα πρέπει ένα δημοκρατικό κράτος να σέβεται την ελευθερία του τύπου. Το ίδιο ασφαλώς επιθυμεί και η Φιλανδία να τηρούνται οι συνθήκες. σημαντικό όμως να υπάρχει σωστή διάδοση ειδήσεων και όλοι να καταπολεμούμε τα fake news, τις ψευδεί ειδήσει. Στη συνέχεια. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσει για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία και εδώ φυσικά το ερώτημα αυτό είναι πολύ εύστοχο. Αυτά που έχουμε αποφασίσει θα πρέπει να εφαρμοστούν και αυτό θα κληθούμε να το συζητήσουμε και στο Συμβούλιο είναι σημαντικό να αξιοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, αυτά από πλευρά μου και τώρα λέει ο Πρόεδρος, η Υπουργό ο Ισάλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις ε, ερωτήσεις σας, την κυρία Μέτσολα, την Ιντφέλτ, Ρασίνη και τους υπόλοιπους. Να ξεκινήσω με τα θέματα ασύλου, σε ό,τι αφορά το κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε αν θέλουμε τελικά να έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από το σημερινό σύστημα. Σε ό,τι αφορά αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά αντιμετώπιση ε, εξαιρετικών μεταναστευτικών ορών. Και όλοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κοινών κανόνων. Και όπως ξέρετε, αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Τώρα λοιπόν είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στου κοινού στόχους. χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη και μια ατμόσφαιρα συνεργασία μεταξύ των κρατών μέλων. Θα πρέπει να κατανοήσουμε με καλύτερο τρόπο του περιορισμού που επιβάλλουν κάποιε εθνικέ καταστάσει. Η Φιλανδική Προεδρία πιστεύει ότι θα πρέπει τα πρακτικά αυτά ζητήματα να τα απαντήσουμε με πρακτικό τρόπο σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια, αναμένοντα ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όταν θα γίνει αυτή η γενική συζήτηση, τότε μπορούμε να κοιτάξουμε και τι συγκεκριμένε λύσει, όπω για παράδειγμα τι διαδικασίε για τα εντάλματα κτλ. Και τα συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα του ποιο θα πάει πού. Η Φιλανδική λοιπόν Προεδρία θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό όσο πιο πολύ γίνεται με το νέο Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα καθοδηγήσουμε τις συζητήσεις για να θέσουμε τα θεμέλια της ε, νέας Επιτροπής και της νέας Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι σαφές, άλλωστε, ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί, το οποίο θα επιτρέψει τη σωστή λειτουργία του συστήματο ε, διάσωση στην Μεσόγειο. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στην ε, ιδέα τη κοινή ευθύνη και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση. Είμαστε όλοι μαζί μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απολύτω απαραίτητο να υπάρχει ένα νέο σύστημα ασύλου το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί γενικά το σύστημα και να επιτροθούμε συγκεκριμένα και στη Μεσόγειο. θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση στη Μεσόγειο με, σε προσωρινό επίπεδο με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Και έχουμε μία έκθεση με τα μη δεσμευτικά στοιχεία του 2019, αλλά θα πρέπει να βρούμε και μία πιο μακροπρόθεσμη ρύθμιση η Επιτροπή θα συντονίσει την δράση αυτή και τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν σε αθλαντική βάση. Η Φιλανδική Προεδρία θα υποστηρίξει φυσικά όλη τη δικασία. Ο αριθμός των πνιγμών στη Μεσόγειο έχει μειωθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ο κόσμος χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να φτάσει στην Ευρώπη θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι θάνατοι στη Μεσόγειο, να μηδενιστούν. Και αυτό θα το πετύχουμε μειώνοντα το κίνητρο του τράφικινγκ, τη εμπορία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την αρχή τη χώρα προέλευση, για να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμο, ε, μάλλον να κοιτάξουμε και τι χώρε προέλευση. προκειμένου ο κόσμο να μπορεί να μείνει στη χώρα του, να μην χρειάζεται να φύγει. Και η Λιβύη προφανώ θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από την διεθνή κοινότητα, γιατί είναι σημαντικό για τους μετανάστες να ξέρουν τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά και η Λιβύη θα πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Έχουμε λοιπόν μία σειρά χωρών που είναι διαθέσιμες να συνεργαστούν για να αποφευθούν συζητήσεις, ε, αποφάσεις ad hoc σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο και όσα συμβαίνουν εκεί. Να σας ευχαριστήσω και για την ερώτηση αυτή που κάνατε. Η Φιλανδία θα εξασφαλίσει ότι θα αναπτυχθούν παρατέρω εξωτερικά μέσα για να υπάρχει διαχείριση της μετανάστευσης σε πνεύμα συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και όλη την βαθύτερη αιτία για τη μετανάστευση. Αν θέλουμε λοιπόν να διαχειριστούμε το θέμα της μετανάστευσης και να βελτιώσουμε την κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρειαζόμαστε σταθερότητα στη Λιβύη. Αυτό προφανώς δεν είναι κάτι το απλό και το μονοδιάστατο. Θα πρέπει να το προσεγγίσουμε από διάφορες πολιτικές οπτικές γωνίες. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στο λαό. Και η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να δράσει συντονισμένα για να υπάρξει σταθεροποίηση της κατάστασης. Η Φιλανδική Προεδρία εκτιμά τη δουλειά που έχει γίνει από την ε, του ΟΗΕ στη Λιβύη και στις γειτονικέ γειτονικές χώρες. Και καλό θα ήταν να συμμετέχουν όσο πιο πολλά κράτη-μέλη γίνεται για την επανεκατάσταση των προσφύγων που διασώζονται στη Μεσόγειο και προέρχονται από τη Λιβύη. Κατά τη Φιλανδική Προεδρία, επίσης, θα εξετάσουμε και το θέμα της πολιτικής επιστροφών για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. μια τευρημένη ενδεχομένως εντολή για την Frontex. Θα κοιτάξουμε επίσης και την πολιτική για τις θεωρήσεις και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η σχέση με τις τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τις επιστροφές συγκεκριμένα. Πιστεύουμε, δε, ότι οι πιο αποτελεσματικές επιστροφές είναι οι βιώσιμες επιστροφές. Και εξετάζουμε την δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μηχανισμών στον τομέα αυτό. Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίπελ. Συμφωνώ ιδιαίτερα ότι όταν μιλάμε για εσωτερική ασφάλεια, φτάνουν πια οι αποφάσεις και τα λόγια. Τώρα χρειαζόμαστε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Για παράδειγμα, μιλάμε για την ασφάλεια στον τομέα 5G, για την ασφάλεια, την ασφάλεια δικτύων. Η παγκόσμια κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου, Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με το 5G. Θα είναι τεράστια η αύξηση των δεδομένων που θα μεταβιβάζονται και θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί αντίστοιχα και η ασφάλεια των δικτύων. Η ασφάλεια των δεδομένων θα αποτελέσει θέμα όλο και πιο σημαντικό όσο περνάει ο χρόνος. Και στις συζητήσεις με τους εταίρους μας το θέμα αυτό πάντα μπαίνει στην ατζέντα. Θα αντιμετωπίσουμε επίσης και προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του δικαίου, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ανάπτυξη του 5G, θα είναι όλο και πιο δύσκολο για τις αρχές επιβόλης του νόμου να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα, γιατί τα δίκτυα 5G και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν ένα θέμα το οποίο επηρεάζει όλες τις πολιτικές γιατί το 5G θα αποτελέσει την τραχοκακαλιά των τηλεπικοινωνιών για το μέλλον και αυτό θα έχει α, επιπτώσεις και στην εσωτερική αγορά, στην ενέργεια, στη βιομηχανία. Θα υπάρχουν λοιπόν θέματα διαχείρισης κινδύνου τα οποία θα ανακύψουν από τη γενιά αυτή. Θα ενέχουν κινδύνους, ε, ευαισθησίες, τις οποίες θα κληθούμε να τις διαχειριστούμε. Και αν μου επιτρέπετε να πω και εν συντομία το εξής. Το θέμα κοινωνική συνοχή, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Φιλανδική Προεδρία, θα το προωθήσουμε ενεργά και δεν μιλάμε μόνο για ενσωμάτωση και ένταξη των ανθρώπων από το εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε και για ένταξη των ανθρώπων που είναι ήδη μέλη και τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μιλάμε για κράτη-μέλη, την ευρωπαϊκή κοινωνία για θέματα κοινωνική ασφάλεια, για θέματα εκπαίδευση. Όλα αυτά μα απασχολούν ιδιαίτερω και πιστεύουμε ότι σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να εξετάσουμε τη συνοχή. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Αν ολοκληρώσατε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, λοιπόν, θα κάνουμε το εξή. Πρώτον, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ε, μελών που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σας πω ποιοι Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους. Όχι με τη σειρά που θα διαβάσω τα ονόματα, γιατί θα προσπαθήσω ως πρόεδρος να διατηρήσω κάποια ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Θα κλείσει ο κατάλογος, αφού τον διαβάσω. Είναι τουλάχιστον 30 τα μέλη που ζητούν να μιλήσουν. καθώς θα σας αναγνώσω τα ονόματα, παρακαλώ να επιδείξετε την ίδια πειθαρχία που επέδειξαν και οι δύο υπουργοί μας εδώ. Για να προσπαθήσετε να τηρήσετε το ένα λεπτό σας. Αλλιώς δεν θα προκάνουμε. Στις 11 έχουμε προγραμματίσει παρουσίαση πεπραγμένων της Europol από την εκτελεστική διευθύντρια, την κυρία Ντεμπόλ. Στις 11 η ώρα. Ακόμα και αν περάσουμε το χρόνο που έχουμε αφιερώσει στην, ε, Λανδική, ε, στην ε, Φιλανδική Προεδρία, συγγνώμη, είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, διαβάζω τα ονόματα. Hidvegi, Mrs. Jaroka, Mrs. Keller, Mrs. Donath, Mrs. Purik, Mrs. Reintke, Mrs. Colin Osterle,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 Ωραία. Κυρία Μπιόρκ, συγγνώμη, δεν το είπα σωστά το όνομά σα, αλλά ήσασταν εγγεγραμμένοι. Ναι. Άλλος. Ε? And? Ε? Okay, I'm I'm get started then. Αρχίζουμε. Όπως σας είπα, θα προσπαθήσω να τηρήσω μια ισορροπία ανάμεσα στις ομάδε. Ένα λεπτό, μην ξεπερνάτε το λεπτό σας. Και μην με κάνετε να χρησιμοποιήσω το σφυράκι. Ο κύριος Χίτιμπεγγι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, είμαι από την Ουγγαρία, λέει ο κύριος Χίτιμπεγγι. Συγχαρητήρια, είναι φιλόδοξα τα σχέδιά σας και συγχαρητήρια για την Προεδρία. Μιλήσαμε για προκλήσεις. Θα ήθελα να σας αναφέρω μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες και πρόκληση, που είναι η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και συνδέεται άμεσα με την λαθρέα μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων. Χαιρετίζω τις προτεραιότητές σας που μιλάτε για συλλογική προστασία και συνολική των πολιτών. Όμως η απάντηση κατά την άποψή μας δεν είναι στη συλλογική διαχείριση της μετανάστευσης. Χρειαζόμαστε σφαιρικά να καταπολεμήσουμε τη λαθρέα μετανάστευση, δηλαδή να καταπολεμήσουμε και το τράφικινγκ και την λαθρέα μετακίνηση, τη διακίνηση ε, προσώπων, οι οποίοι πέφτουν θύματα εκείνων ε, που τους εκμεταλλεύονται και ορισμένοι ε, μπορεί να το κάνουν εσκεμένα ή όχι. Ερωτώ λοιπόν πώς προτίθεται η Προεδρία να βοηθήσει για να δημιουργηθούν πλατφόρμες αποβίβασης σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 28-29 Ιουνίου για να καταπολεμήσουμε ε, τους λαθροδιακινητές και να τους στέλνουμε πίσω αντί να τους φέρνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους μετανάστες γιατί αυτό θα, αποτελέσει και μια αποτροπή της έλευσης τους εδώ στην Ευρώπη. Ε, κύριε Πούρεκ, σας. Αγαπητοί Υπουργοί, ε, σας ευχαριστώ. Αγαπητές Υπουργοί, μάλλον θέλω να θέσω δύο ζητήματα εδώ, ενδοοικογενειακή βία και έμφυλη βία. Είμαι εισηγήτρια για την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Χαίρομαι που η Φιλανδία ήταν από τις πρώτες χώρες που την υπέγραψε και πολύ σύντομα στη συνέχεια την κύρωση. Ε, όμως γιατί Ρουμανία τη Φιλανδία και την Κροατία, το τρίο, δεν έχει αναφερθεί ε, σε αυτό το θέμα ρητά και ε, το θέμα εκρεμεί και περιμένουμε όλοι ε, να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η καταπολέμηση της υγείας κατά των γυναικών δεν μπορεί να περιμένει όμως και να εκρεμεί. Ερωτώ, τι προτίθεται ακριβώς να κάνει η Φιλανδική Προεδρία σχετικά. ακόμα και αν δεν αναφέρετε ρητά το θέμα στα επίσημα έγγραφα της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ κυρία Κέλε. Κελέχ, Φαμπιέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, το δικό μου θέμα αφορά ε, το κοινό καθεστώς ευρωπαϊκού ασύλου. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε νομοθετική δέσμη από το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ε, θέση και εντολή διαπραγματευτική για όλα τα θέματα. Αυτό αφορά ε, τη διεκπαιρέωση των αιτημάτων ε, ασύλου, των αιτήσεων και την όλη διαδικασία υποδοχής και φιλοξενίας. Κυρίες Υπουργοί, η Φινανδική Προεδρία έχει τη φιλοδοξία να προωθήσει αυτά τα θέματα και να προτείνει και χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των κειμένων αυτού του πακέτου για το άσυλο. Επιτρέψτε μου να σας ερωτήσω ιδιαίτερα για το θέμα ε, του κανονισμού του Δουβλίνου που διέπει το άσυλο. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα να μας δώσετε και μια μέθοδο για να προχωρήσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρέτκε, για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Να σας ρωτήσω μετά από τους ε, δύο συναδέλφους, η... είναι μεν προτεραιότητα η προσχώρηση στη Σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά οδηγία κατά της έμφυλης βίας από το Συμβουλίο. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε. Η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει εκφράσει την επιθυμία να κινηθεί και η Φιλανδική Προεδρία προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Καπτίνο, κυρία Καπτίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σωστά είπατε πως υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη και στην Ιταλία υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δυσκολίες με τα θέματα ασύλου. Βέβαια, το η δέσμη μέτρων για το άσυλο έχει δημοσιευτεί εδώ και τρία χρόνια, όμως Σε ό,τι αφορά το στάδιο της έγκρισης, ε, οι ταχύτητες ε, στο Συμβούλιο διαφέρουν. Από τα τέλη Ιουνίου πέρυσι έχουν... Διάφορα κράτη-μέλη έχουν μπλοκάρει το θέμα και δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απομονωθούν ορισμένα κράτη-μέλη και να μείνουν μόνα τους στην προσπάθεια να διαχειριστούν την ε, πρόσφυγη και μεταναστευτική κρίση. Αυτό έχει οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, με τη διακίνηση ανθρώπων κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Φιλανδική Προεδρία αν είναι ε, προτεραιότητά του στο θέμα αυτό και αν θα είναι σε θέση να μας δώσει μία επίσημη θέση για τη δέσμη μέτρων για το άσυλο και αν ε, μας δώσει αποτελέσματα για αυτό το πολύ ουσιαστικό πραγματικό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λακοντίνσκι εκ μέρους της ομάδας ECR. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, τα, το PNR, τα ονόματα των επιβατών. Μας εξέπληξε η παρουσίαση της ε, Προεδρίας σας που θεωρεί προτεραιότητα τη διεύρυνση του PNR και σε άλλα μέσα και πρόσφατα το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η παρόμοια συμφωνία με τον Καναδά παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς πώς μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα αυτά, τι, τι, έχετε να μας πείτε. Έπειτα, σχετικά με το κράτος δικαίου. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της αναθεώρησης αυτής. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή τι, τι θα αναθεωρήσετε θα εξετάσετε τα συστήματα δικαιοσύνης και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά. Εμείς θα θέλαμε φυσικά να δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά ας τα αφήσω το θέμα εκεί. Επίσης, τι ε, άποψη έχετε για το, ε, το την πολιτική διάσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Κολένα Σταρλέ, στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τη εγκληματικότητα μιλήσατε για την πρόθεσή σας να διευρύνετε το πεδίο εφαρμογή του PNR, τα στοιχεία δεδομένων επιβατών, και σε άλλα μέσα μεταφοράς, δηλαδή και στην αψιπλοεία αλλά και στα ε, διεθνή τρένα υψηλή ταχύτητας. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2015 έγινε μια γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, απάντησε ότι δεν ε, προτίθεται να κάνει μελέτες για το σιδηρόδρομο. Εσείς από ό,τι φαίνεται θέλετε να το κάνετε προτεραιότητα της Προεδρίας σας. Το έχετε θέσει υπόψη στους εκπροσώπους των κρατών μελών και της Κομισιόν και αν ναι, έχετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για τα μέσα αυτά μεταφοράς ή ακόμα και για το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους, ε, τις υπουργούς να σας ευχαριστώ για την επισκεψή σας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θέτουμε τις προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες με τέτοια βασικά ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Σε αυτά συγκαταλέγεται και η μετανάστευση. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιοι απαράδεκτων καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο, όπου οι μετανάστες ε, ξεμένουν ε, σε τέτοιες καταστάσεις στη Μεσόγειο, στο Ιόνιο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μένουν στη θάλασσα. Θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα, θα πρέπει να προτείνουμε μέτρα ασφάλειας τα οποία συγκαταλέγονται και αναφέρονται μάλιστα και στην ε, συνθήκη του Δουβλίνου, την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν τι προτεραιότητέ μα και θα πιστεύετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε τέτοιε αποφάσει. Θα μπορούσαμε σύμφωνα με τη συνθήκη να προχωρήσουμε με ειδική πλειοψηφία. Στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που μας μπλοκάρουν. Αλλά όπως και αν το κάνουμε υπάρχουν θέματα στα οποία δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε αλληλεγγύη στα διάφορα θεσμικά όργανα και μεταξύ κρατών μελών, όπως το άρθρο 80. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, να προσαρμόσετε τις ερωτήσεις σας στο ένα λεπτό που έχετε στη διάθεσή σας. Η επόμενη βρυδιά από το The Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω την Φιλανδική Προεδρία σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε και σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου που έχουν θέσει ω προτεραιότητα, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά επίση. Αναφέρθηκε και το θέμα του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωση. Ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η τοποθέτηση τη φιλανδική Προεδρίας, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση του πλουραλισμού του τύπου με το κράτος δικαίου, ιδιαίτερα σε τέτοιε χώρε όπου υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία χωρί πλουραλισμό στο μέσα ενημέρωση. Και μιλάω για την Ουγγαρία και μιλάμε για τι διαδικασίε του άρθρου 7. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πληροφορίε που μα δώσατε. Σα παρακαλώ όμω, για να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε ό,τι αφορά την ακρόαση αυτή ενώπιον του Συμβουλίου, πότε θα λάβει χώρα, τι σκοπεύετε να κάνετε και πώς θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτά. Λίγο πιο συγκεκριμένα από αυτά που μα είπατε προηγουμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κ. Μακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις, κυρίες Υπουργοί. Δύο ερωτήσει να κάνω. Προφανώ ε, η αλλαγή του, κύκλου, του κλίματος αποτελεί προτεραιότητα για τη Φλανδική ε, Προεδρία και το συμφωνώ με αυτό, γιατί συνεπάγεται και μετανάστευση. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε προστασία από την αλλαγή του κλίματος. Δεν έχουν δικαίωμα να θεωρούνται πρόσφυγες, δεν απολαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα τέτοια, άλλη τέτοια προστασία στα κρατη Τι επισκοπεύει λοιπόν να κάνει η Φιλανδική Προεδρία και για την αλλαγή του κλίματος φυσικά, αλλά και για τους ανθρώπους που μεταναστεύουν για λόγους αλλαγής του κλίματος. Και φαντάζομαι ότι είπατε τον Μπόρις Τζόνσον που έχασε με τρεμβευτικό τρόπο στο, στην καταβουλή. Α, παρ' όλα αυτά όμως βγαίνει και τετρανώνει την πρόοδο που έχει πετύχει στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας εσείς που τα ξέρετε, έχει πετύχει οποιαδήποτε νίκη, ο Μπόρις έχει κάνει οποιαδήποτε πρόοδο ή μήπως λέει ότι θέλει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μιλήσω αγγλικά, αλλά θέλω να χαιρετήσω στα σουηδικά. Τρία πράγματα έχω να πω για το κράτος δικαίου. Πιστεύω ότι έχετε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο. Να κάνω μια ερώτηση όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση των ΜΚΟ και την ε, αλληλεγγύη προς τους ε, πρόσφυγες και τη μείωση της ε, κοινωνίας των πολιτών. Κατά δεύτερον, το θέμα της βίας βάση του φύλου. Αυτό αποτελεί προφανώς θέμα και αντικείμενο και της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Και τέλος, είμαι η συγγήτρια για τον φάκελο για το θέμα της επανεγκατάστασης από πλευράς του Κοινοβουλίου. Το Έχουμε προχωρήσει το θέμα αυτό σε ένα θέμα ανθρωπιστικό το οποίο δεν έχει βάση στην αιρεσιμότητα. Θέλω λοιπόν να προχωρήσουμε το θέμα αυτό με τη Φιλανδική Προεδρία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αποτελεί ε, έναν από τους μοναδικούς νόμιμους και ασφαλείς τρόπους για τους μετανάστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιάροκα για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Όχι μόνο για το πώς θα σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση, αλλά και το πώς τα άτομα αυτά μπορούν να επιστραφούν και πώς να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πώς να βοηθήσουμε και την Αφρική και τις άλλες περιοχές από τις οποίες φεύγει ο κόσμος. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν έχουμε σχετική τεχνογνωσία και στην Ευρώπη είναι πολύ λίγε αυτέ οι καλέ πρακτικέ ό,τι αφορά τη μείωση τη φτώχεια. Το 2011 η Ουγγρική Προεδρία εισήγαγε ένα σχέδιο για 43 εκατομμύρια τότε ανθρώπου, γιατί είναι πάρα πολύ η φτωχοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί είναι από μειωτικέ ομάδες και πολλοί από είναι Ρωμά. Χρειαζόμαστε λοιπόν υγειονομικές εγκαταστάσεις, νερό, δεν έχουν ε, μπάνια, δεν έχουν τρόφιμα το πιο βασικό. Άρα πιστεύω ότι η Φιλανδική Προεδρία που το 2000 ήταν τόσο προοδευτική σε θέματα Ρωμά θα πρέπει να δείξει εκ νέου την τόλμη και το θάρρος της για να προχωρήσει το θέμα αυτό παράλληλα με τα οικονομικά προγράμματα για την ε, Φιλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ, κύριε Μωράης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργοί. Να σταθώ λίγο στο θέμα για την στήριξη στην υπηρεσία ασύλου. Κατανοώ την αγανάκτηση πολλών συναδέλφων σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Να πω όμως ότι, όπως είπε ο συνάδελφος Μπαρτόλομη, εσείς ε, έχοντας την Προεδρία έχετε και το ρόλο του διαμεσολαβητή. Γι' αυτό λοιπόν οφείλετε να προσπαθήσετε ε, να πιέσετε, διότι η ενισχυμένη πλειοψηφία είναι στις συνθήκες, δεν είναι κάτι που είναι απλά επιθυμητό. Δεν γίνεται λοιπόν το Συμβούλιο να συνεχίσει να μπλοκάρει πράγματα μόνο και μόνο επειδή έτσι θέλει. Μετά υπέρχεται η αδράνεια. Γι' αυτό λοιπόν ε, η πρότασή σας ε, περί είναι καλή, είναι έξυπνη, όμως φοβάμαι πως τα ίδια προβλήματα θα προκύψουν και θα προκύπτουν ξανά και ξανά. Έπειτα, διαβάσαμε το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαδικασία ασύλου, για το Δουβλίνο ε, και εσείς έχετε κάποιες παραπάνω, παραπάνω πληροφορίες για το τι θα παρουσιάσει, διότι στην Μάλτα, στην ε, Ιταλία στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σιμέτσκα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι τα όσα είπατε για, για το κράτος δικαίου, αλλά έχω μια ερώτηση σχετικά με την εργαλειοθήκη, την οποία θα συζητήσουμε τους ερχόμενους μήνες. Αναφερθήκατε στα συστατικά στοιχεία αυτής της εργαλειοθήκης και ότι θα διαδραματίσει ρόλο διευκολυντή διαλόγου. Αναφερθήκατε επίσης στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Όμως, τι συμβαίνει με τα διορθωτικά μέτρα και μας μιλήσατε μεν για τη σύνδεση της χρηματοδότησης με τις ευρωπαϊκές αξίες και τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για κυρώσεις. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός ε, διορθωτικού μηχανισμού διορθωτικών μέτρων πέρα από εκείνων που διαθέτουμε ήδη. Ε, αναφέρομαι φυσικά στην περίπτωση που το άρθρο 7 δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα, που έχουμε δύο γυναίκε υπουργού εδώ, αλλά και σε τέτοιε κρίσιμε ε, θέσει ε, που χρειάζονται φεμινίστριες. Αυτό σπάνια συμβαίνει σε άλλα κρατημέλη και χαίρομαι ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ. Αναφέρατε την αποφασιστικότητά σα για το άρθρο 7. Αυτό το έφεραν διάφοροι βουλευτέ. Είπατε ότι θέλετε διάλογο με το Κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την έκρηση τη έκθεση για την Ουγγαρία, ή το Κοινοβούλιο δεν είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη θέση της και την έκθεση του στην, ε, στο Συμβούλιο και για την Πολωνία. Και έτσι λοιπόν η έλλειψη της άποψης του Κοινοβουλίου αποτελεί ένα μεγάλο αρνητικό σημείο στην όλη διαδικασία αυτή. Θα μπορέσει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην Ακρόαση και κάτι άλλο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, αλλά μιλάμε για την ε, υποψηφιότητα για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικέ απόψει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σήμερα, λοιπόν, η υποψηφία ε, τη Γαλλία έχει πάρει άλλη θέση. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο υποψήφιος. Θα προχωρήσει λοιπόν το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάλη. Όχι, θα συντήσατε το λόγο πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρο. Μάλιστα θα σα διαγράψω. Ο Σαχαλέχος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργοί, εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Να σταθώ σε κάποια επιμέρους θέματα. Πρώτον, την ε, πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Υπάρχουν στη διάθεση της Φιλανδικής Προεδρίας κάποια νέα στοιχεία έτσι ώστε να προσθεθούν στην στρατηγική πρόληψης. Έπειτα, η Φιλανδική Προεδρία πώς έχει αξιολογήσει την κατάσταση της δικαστικής συνεργασίας στην Ένωση. Θεωρείτε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θεωρείτε πως η εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα μπορεί να βοηθήσει, διότι ο τομέας της δικαστικής συνεργασίας είναι πραγματικά σημαντικός, ακρογωνίως λήθος. Και χρειάζεται λοιπόν ε, να τον ενισχύσουμε έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδος στην ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην Επιτροπή μας να μας παρουσιάσετε ε, το πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Όταν ήρθα στην Ευρώπη, ήμουν προσφυγόπουλο και για μένα η Ευρώπη ήταν ο η μόνη σωτηρία και δυστυχώς ο μόνος τρόπος για να φτάσω στην Ευρώπη ήταν παράνομος. Τώρα υπάρχουν νόμιμε, νόμιμοι τρόποι να φτάσει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε όμως ότι η παρανομία συνεχίζει και επεκτείνεται και ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πέφτουν θύματα ε, διακίνησης, εκμετάλλευσης. Μιλάμε τώρα για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε για ένα από τα πιο μεγάλα σε έκταση εγκλήματα. Και γίνεται σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Επίσης, πολλές γυναίκες χάνουν τη ζωή τους. Περίπου 7 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ε, ε, επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τι θα κάνετε για να πιέσετε τα υπόλοιπα κράτη να το πράξουν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρέιερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητές Υπουργοί, η ερώτησή μου έχει να κάνει με τον κανονισμό για την ε, ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Είχαμε την, έκθεση, στην, την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο είχε να προστατεύσει τους πολίτες από το να τους ε, παρακολουθούν στο διαδίκτυο, να παρακολουθούν τις κινήσεις τους. Όμως βλέπω ότι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν είναι τόσο ισχυρές σήμερα η Προεδρία σας θα πιέσει επιτέλους το Συμβούλιο να λάβει μία επίσημη θέση. Ξέρω πως αυτό θα συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, όμως εσείς ως εκπρόσωποι της Προεδρίας μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόζενμπεργκ. Πρόεδρε, Κυρίες Υπουργοί, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Παρακολούθησα με πολύ προσοχή τις θέσεις σας απέναντι στην ανάγκη μεταρρύθμισης του Δουβλίνου, της πολιτικής των επιστροφών, τους πρακτικούς τρόπους που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν άκουσα όμως την θέση της Φιλανδικής Προεδρίας σε σχέση με εκείνες τις χώρες που δεν δέχονται να υποδεχθούν τους πρόσφυγες που με δημοκρατικές αποφάσεις έχουμε αποφασίσει, τι σκέφτεστε να κάνετε αν πρόκειται να προτείνετε οικονομικές κυρώσεις ή μια άλλη πολιτική διότι οι συμπατριώτες μου στην Ελλάδα που έχουμε υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος αμφισβητούν την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία θεωρούν ότι μόνο στα έγγραφα υπάρχει και όχι με πρακτικό τρόπο σε ανταπόκριση όλων των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω εδώ τον κύριο Παπαδάκη. Α, εδώ είναι, μάλιστα. Έχετε το λόγο, κύριε Παπαδάκη. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, για το προσφυγικό θα μιλήσω. Στη Λέσβο αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα είναι για 3.000 το hot spot και διαμένουν πάνω από 11.000. Στη Σάμο η χωρητικότητα 700 ζουν σχεδόν 5.000. Στα άλλα hot spot διπλάσιοι και τριπλάσιοι και αυτή την ώρα που μιλάμε 65.000 μετακινούνται εσωτερικά στην Τουρκία και είναι ε, αρκετά πιθανό κάποιοι από αυτοί να καταλήξουν πάλι στα νησιά τα ελληνικά. Είναι αδιέξοδος ο εγκλωβισμός με βάση την συμφωνία, την απαράδεκτη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας που κάνει αβίωτη την κατάσταση και για τους πρόσφυγες και για τους νησιώτες στην Ελλάδα. Να κλείσουν τώρα τα απαράδεκτα hot spot, να δημιουργηθούν ανθρώπινες αξιοπρεπείς Υποδομέ φιλοξενίας στις χώρες τελικού προορισμού. Και θέτουμε το εξή. Η κυβέρνηση τη Νέας Δημοκρατίας, η καινούρια, ε, προωθεί την κατάργηση της δευτεροβάθμιας εξέτασης ασύλου. Πρόκειται για απαράδεκτη κίνηση που ε, καταργεί στοιχειώδη δικαιώματα και ελευθερίες και θα θέλαμε την γνώμη των δύο Υπουργών. Ευχαριστώ. Thank you. Last minute. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω την ε, Φιλανδική Προεδρία γιατί ήταν πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει ως τώρα και είμαι ο εισηγητής για το θέμα του πολιτικού δημοσιονομικού προϋπολογισμού και σε ό,τι αφορά το θέμα του κράτους δικαίου και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρώπων με αναπηρία θα ήθελα να αναφέρω σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τις Αναφορές έχει λάβει διάφορες τέτοιες επιστολές και από ό,τι φαίνεται στη Φιλανδία Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ε, ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση που τελικά οι ανάπηροι δεν έχουν πρόσβαση επαρκή τουλάχιστον σε θέματα λήψη ε, λήψης αποφάσεων ή α, θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω λοιπόν να σας ε, απευθύνω το εξή ερώτημα, κυρία Υπουργέ. Τι μέτρα θα πάρει η Προεδρία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αναπήρων και συγκεκριμένα η Φιλανδία θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ελέγξει κατά πόσον η εφαρμογή των οδηγιών είναι αντίθετη με την σύμβαση του ΟΗΕ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν τώρα 7 λεπτά για την κάθε Υπουργό για να απαντήσει. Έχουμε και τον ε, ε, διευθυντή της Europol, ο οποίος περιμένει. Θα σας ζητήσω λοιπόν να είσαστε σύντομες, αλλά μας αποδείξετε και στην προηγούμενη, στον προηγούμενο γύρο ότι είσαστε πολύ συνοπτικές. Ε. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να απαντήσετε στις ερωτήσεις της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο πολλές ερωτήσεις γίνεται. Γιατί ακούσαμε πολλές και καλές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών και την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες. Και όλοι μας θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό, γιατί είναι απαράδεκτο. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε τις χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση να την επικυρώσουν. Πέραν τούτου, ως ε, Προεδρία του Συμβουλίου θα θέλαμε να προσπαθήσουμε να ενταχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύμβαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντως έχει μία γνωματοδίση και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουμε σχετική απόφαση. Τα δικαιώματα λοιπόν των θυμάτων θα πρέπει να ενισχυθούν και ως Προεδρία θα πρέπει να θέξουμε το θέμα αυτό στους κόλπους του Συμβουλίου. Το θέμα της προστασίας των θυμάτων δηλαδή. Θα θέλαμε να τονίσουμε επίσης ότι η σχετική οδηγία για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών θα πρέπει να τονιστεί. Ο ρόλος λοιπόν των γυναικών είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και χαιρόμαστε που η μελλοντική πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, φροντίζει και επιθυμεί να υπάρχει ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην μελλοντική επιτροπή. Γιατί το θέμα είναι και μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την ίση εκπροσώπηση των φύλων. Επίσης, ε, αναφέρθηκαν κάποια άλλα σημεία. Αυτό το Justice Scoreboard, αυτό τον πίνακα αξιολόγηση στο θέμα των δικαιοσύνης. Ε, θέλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό γιατί αποτελεί ένα ακόμα μέσο για την τήρηση του κράτους δικαίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την Πολωνία και την Ουγγαρία. ζητήσατε πιο συγκεκριμένε πληροφορίε σε ό,τι αφορά το follow-up. Το Συμβούλιο λοιπόν προβλέπει μια πρώτη α, ακρόαση το Σεπτέμβριο με την Ουγγαρία, μέσα στο μήνα δηλαδή. Και θα δώσουμε την ευκαιρία στην Ουγγαρία να σχολιάσει την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Υπουργό του Περάιν, ο οποίο είναι επικεφαλή του Συμβουλίου, θα συναντηθεί σήμερα και με εκπρόσωπο της Επιτροπής σας για να ακουστεί και η δική σας φωνή. Σε ό,τι αφορά την Πολωνία, η έκθεση της Κομισιόν εξετάστηκε στο Συμβούλιο τον Ιούλιο, το Συμβούλιο το Ιούνιο έλαβε σημαντικές ε, πληροφορίες και εξέδωσε σημαντικές πληροφορίες, μία ενημέρωση. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Ζητήσατε και συγκεκριμένες, συγκεκριμένα στοιχεία για τις ε, επερχόμενες ακροάσεις. Προφανώς θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαρθρωμένη διαδικασία. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα λάβει η χώρα η ακρόαση για την Ουγγαρία σε αυτό που είπε η κυρία Μπιόρκ. Και σας ευχαριστώ παρεμπιπτόντως για την ερώτηση που μου κάνατε για την διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Είμαστε μια κοινότητα αξιών, το τονίζω αυτό. Και ω τέτοια πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους σε ό,τι αφορά θέματα διάκριση, διακριτική μεταχείριση ε, κατά τον Ρωμά, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Εδώ να τονίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η αρχή της αντιμετώπισης των ανθρώπων και αυτό θα το προωθήσουμε ως Προεδρία. Η διακριτική λοιπόν μεταχείριση αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα, εξακολουθεί να υπάρχει, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα. Μόνο με βιώσιμότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά μακροπρόθεσμα. Και το θέμα της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης αφορά και τις μειον, μειονότητες. Να ευχαριστήσω σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ταχθεί ενεργά υπέρ των δικαιωμάτων του Ρωμά. και τη συμμετοχή της Ρουμανίας για την καταπολέμηση των ε, μέτρων που είναι επιθετικά κατά τον Ρωμά. Αναφέρατε επίσης το ρόλο του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου, είναι κάτι το οποίο συζητιέται και συζητήθηκε ε, γενικότερα όταν αναλάβαμε την Προεδρία τα κράτη-μέλη ζήτησαν ε, στην αρχή της ακρόασης να έχει επαφές η Προεδρία με το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σκοπεύουμε να βρούμε μια λύση το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο. Επισήμως δεν έχουν γίνει οποιασδήποτε ανακοινώσει. Δεν έχει αποσύρει κανείς την υποψηφιότητά του. Είναι σημαντικό όμως να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Ελπίζω το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά την διακίνηση ανθρώπων τώρα. Φυσικά η διακίνηση ανθρώπων είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από τις συνθήκες. θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την υποστήριξη των θυμάτων. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για την ασφάλεια των δεδομένων, εδώ θέλουμε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα του e-privacy. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα εσείς, Υπουργέ, όχι άλλο, για τα επόμενα 7 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω και σας ε, Πρόεδρε, και όλους τους ε, βουλευτές για τις καταπληκτικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ και την κυρία Χένιξον. Το PNR. Κοιτάξτε, οι τρομοκράτες και οι κλιματίες δεν ταξιδεύουν μόνο με αεροπλάνα, χρησιμοποιούν και άλλα μέσα μεταφοράς για να προλάβουμε την τρομοκρατία και τη σοβαρή εγκληματικότητα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, να εξετάσουμε τα πιθανά πλεονεκτήματα της επέκτασης του συστήματος PNR και σε άλλα μέσα μεταφοράς. Το Συμβούλιο έχει βγάλει σχετικά συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές και άλλες συνέπειες. Η Φιλανδία δεν αναμένει βραχυπρόθεσμα να εγκριθεί νομοθεσία, αλλά η οδηγία για τα ε, δεδομένα των επιβατών, των PNR, είναι δύσκολη στην εφαρμογή της, στην καθημερινή. Η ευρεία χρήση δεδομένων PNR χρειάζεται ε, ανάλυση ε, και μελέτη αντικτύπου εμπεριστατωμένη πριν εφαρμοστεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να μεταβιβάζονται σήμερα ε, τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και ε, χάνουν ηλεκτρονικής επεξεργασίας και αυτή η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του Δουβλίνου και το πακέτο για το άσυλο, το βασικότερο ζήτημα που χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η Φιλανδία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτή τη δουλειά της μεταρρύθμισης. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και για μια επικοδομητική συνεργασία όλων των κρατών μελών σε ένα τέτοιο πνεύμα σε όλους τους τομείς του ασύλου. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να σταματήσουμε αυτούς τους πνιγμούς στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή δεν τα πάμε καλά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μεταξύ άλλων είναι να βεβαιωθούμε ότι θα μπορούν τα σκάφη και οι βάρκες να ελιμενίζονται και να ε, αποβιβάζουν τον κόσμο γρήγορα. Ε, ε, μπορεί να χρειαστεί προσωρινή λύση, γιατί η μόνιμη λύση θα αργήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθούν όσο γίνεται οι χώρες εκείνες που εθελοντικά ε, θα μοιράζονται αυτό το βάρος. Η Φιλανδία θα κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει αυτή την υπόθεση του Δουβλίνου. Σε ό,τι αφορά τώρα τους επαναπατρισμούς και τις επιστροφές. Η Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου θα φροντίσει να δώσει κίνητρα ή να αναζητήσει κίνητρα για τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να ε, δέχονται εκείνους που επιστρέφουν. Υπάρχουν δυνατότητες στην πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίων και με άλλους τρόπους μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Αυτό πραγματικά έχει δρομολογηθεί. Εθελοντικές επιστροφές είναι και παραμένει ένα ε, ζήτημα κλειδί. Το υποστηρίζουμε και ε, θέλουμε να βεβαινόμαστε ότι είναι βιώσιμες αυτές οι επιστροφές και μόνιμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική. Η εξωτερική εντολή του Frontex δίνει δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως. Για την Ελλάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφήξεις στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία και γνωρίζουμε ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στα νησιά αυτά. Θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την Ελλάδα και οικονομικά και επιχειρησιακά έτσι ε, ώστε να είναι σε θέση τα ελληνικά νησιά να υποδέχονται αυτούς τους μετανάστες. Οι ευάλωτες ομάδες την χάνουν ιδιαίτερη προστασία. Για την καταπολέμηση της, ε, του εξτρεμισμού Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας η Φινλανδία προτίθεται να ε, προωθήσει τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη ε, για να καταπολεμούν την ακραία βία, την εξτρεμιστική βία. Η Φιλανδία ε, θέλει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αναλύσουν τη δυνατότητα πρόληψης της ζωσπαστικοποίησης και της βίαιης συμπεριφοράς. Υπάρχει ένας μηχανισμός ε, συντονιστικός για τη ριζοσπαστικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή, να εργάζεται ε, με ανοιχτό πνεύμα, έτσι ώστε ε, να υπάρξει ένα σύστημα αποτελεσματικό και βιώσιμο. Η Προεδρία θα υποστηρίξει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και φυσικά ενθαρρύνει όλους να συμμετέχουν πλήρως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you so much. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χένριξον ζήτησε λίγο ακόμα χρόνο, 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μπορέσει να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις και θα τον έχει αμέσως τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο αγαπητό Ευρωβουλευτή από τη Φιλανδία ρώτησε, έκανε μια ερώτηση για τα άτομα με αναπηρία. Να απαντήσω λοιπόν ότι φυσικά και θέλουμε να ε, προσπίζουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Η ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να στηρίξουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα κράτη-μέλη. Οφείλουμε λοιπόν να φροντίσουμε να, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι νόμοι. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, τώρα ήρθε η ώρα και για εμάς να δείξουμε την εκτίμησή μας και όπως κάνουμε κάθε εξάμεινο σε αυτήν την Επιτροπή. Να ευχηθούμε λοιπόν στη Φιλανδική Προεδρία κάθε επιτυχία. Αλλά να ευχαριστήσουμε και τις ε, κυρίες Υπουργούς για την ακρίβεια και την ε, λεπτομέρεια που ε, παρουσίασαν σε, ε, κρατώντας ταυτόχρονα το χρόνο αγόρευσης πιστά. Θα ήθελαμε λοιπόν να τις ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να τους ευχηθούμε καλή τύχη στην Προεδρία. και να πω ότι δεν είναι πρώτη φορά που η Φιλανδία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από 20 χρόνια ανέλαβε την Προεδρία για πρώτη φορά και το αποτέλεσμα του εξαμήνου αυτού ήταν το Τάμπερε. Νομίζω όμως ε, πως ε, πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα σε αυτήν την ιστορική στιγμή ως Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνη και Δικαιοσύνης και να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τις κυρίες Υπουργούς, να τους ευχηθούμε καλή τύχη.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

Please, Σας παρακαλώ, καθίστε. Όπως σας είπα και πριν, έχουμε πολλά στην ημερήσια διάταξη και προχωράμε λοιπόν με το επόμενο σημείο της, με μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων των Οργανισμών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ξεκινώντας με την Ευρωπόλ. Έχουμε εδώ την ε, εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ, την Κάτριν ε, Ντεμπόλ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμότατα στην Επιτροπή μας. Και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μία ώρα και 15 λεπτά για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα έχουμε τον ε, συνηθισμένο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές, μετά απαντήσεις και μετά από, τους, από τα μέλη της Επιτροπής. Σας παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε το χρονομιλία σας, διαφορετικά δεν θα προλάβουμε. Επίσης μην ξεχνάτε πως θα μας ενημερώσουν όλοι οι εκτελεστικές, εκτελεστικοί διευθυντές όλων των ε, οργανισμών σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τώρα το λόγο αυτή αμέσως στην Κάτριν Ντεμπόλ για να μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ και τα ευρήματα της πρόσφατα δημοσιευμένης έκθεσης για την κατάσταση με την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπόλ προεδρεύει του δικτύου των εννέα οργανισμών που υπάγονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της κυρίας Ντεμπόλ και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις των συντονιστών. Κυρία Ντεμπόλ, έχετε το λόγο για περίπου 15 λεπτά έτσι ώστε να μπορέσουν οι συντονιστές και τα μέλη της Επιτροπής να σας κάνουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Ευρωπόλ στην, ε, συνεδρίασή σας. Είναι μία από τις Πρώτε συναντήσει τη νέα θητεία. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε πάρα πολύ που μα καλέσατε να σα παρουσιάσουμε το έργο τη Ευρωπόλ. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην Προεδρία ε, του Δικτύου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και θα ε, συνεχίσω καταλήγοντα τα αποτελέσματα και τα ευρήματα σχετικά με την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποστολή της Ευρωπόλη είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη μέσω της πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μετόπων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεγκλήματος δεν είμαστε FBI της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε ε, κάποιον να κάνει έρευνα. Το μόνο που κάνουμε είναι να συντονίζουμε τις έρευνες σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Η Ευρωπόλ θεωρείται ένας έμπιστος εταίρος ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αρχές επιβολής του νόμου και ο οργανισμός μας είναι αξιοσέβαστη αρχή για θέματα στρατηγικής. Η ε, στρατηγική την οποία καταρτίζουμε πολλές φορές και για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και για τα κρατημέλια και για τρίτες χώρες. Η επιχειρησιακή στήριξη είναι κάτι που επίσης προσφέρουμε μέσω του δικτύου μας. Σε όποιον μας το ζητήσει έχουμε μία μεγάλη εργαλειοθήκη, έχουμε μέσα και υπηρεσίε τα οποία προσφέρουμε σε όποιον τα ε, χρειάζεται. Η Ευρωπόλ έχει σκοπό να γίνει το κέντρο δίευλος ε, όλων των ε, πληροφοριών για ποινικά ζητήματα. Αυτό αυτά που μπορεί να ε, επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει η Ευρωπόλ περιγράφονται με λεπτομέρειες στην εντολή λειτουργίας της. Επίσης, η Ευρωπόλ συνδέει τα κράτη-μέλη μεταξύ τους, τους ε, δίνει νέα στοιχεία για να προχωρήσουν οι έρευνες, εγκληματολογικές αναλύσεις και από το 2015 στηρίζουμε τις ε, περισσότερες έρευνες σχετικά με την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, την ε, Κολονία, τη Βαρκελόνη, τη Στοκχόλμη. Πολλές από αυτές τις ε, υποθέσεις που επεξεργαζόμαστε διεξάγονται από κοινού με την Eurojust λόγω του κοινού συμφέροντος και για μια γρήγορη εξέλιξη της υπόθεσης. Παρέχουμε λοιπόν στήριξη στα κράτη-μέλη, παρέχουμε τα εργαλεία και τα μέσα ε, για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα. Τους ε, δίνουμε εργαλεία που σπανίζουν, που δεν έχουν στη διάθεσή του τόσο συχνά οι αρχέ επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα καταπολέμηση ηλεκτρονικού εγκλήματο, κρυπτονομίσματα κτλ. Επίση, όταν προκύπτει ανάγκη, η Ευρωπόλ παρέχει εκτεταμένη στήριξη σε αρχέ των κρατών μελών, για παράδειγμα τη Μάλτα και της Σλοβακίας μετά από τις δολοφονίες του Γιάννη Κούτση και της Δάφνη Καρουάνα στη Μάλτα και τη Σλοβακία των δημοσιογράφων αυτών. Η Ευρωπόλ επίσης είναι ένας αξιόπιστος ε, εταίρος για τα κράτη-μέλη και αυτό φαίνεται από την αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών μας, καθώς και από την ε, γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων τα οποία μοιραζόμαστε. Ε, πέρυσι φτάσαμε το 1,1 εκατομμύρια επιχειρησιακά μηνύματα που ε, λάβαμε και στείλαμε. 77.300 νέες επιχειρησιακές υποθέσεις το 2018. Ένα σύνολο ε, που φτάνει το 66% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πάνω από 1.700 υποθέσεις ε, στην επικράτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασυνοριακές, που στηρίξαμε και πάλι μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2016 και το 2018 ε, στηρίξαμε 620 υποθέσεις τρομοκρατίας. Υπάρχει κέντρο για το κυβερνοέγκλημα, κέντρο για την τρομοκρατία, για το λαθρεμπόριο και κέντρο επιχειρήσεων για το οργανωμένο έγκλημα που καλύπτει και τους άλλους τομείς ε, εγκληματικής δραστηριότητας όπως διακίνηση ναρκωτικών. Οι εγκληματικέ οργανώσει επωφελούνται από την παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στι δευτερογενεί μετακινήσει των ευάλωτων ομάδων, των ομάδων δηλαδή που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα ε, εγκληματιών. Πέρυσι η ασπινική αστυνομία στηρίχθηκε από την Ευρωπόλ για την ε, διάλυση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν ε, διακινώντας ανήλικους από το Μαρόκο στην Ισπανία. Επίσης, στηρίξαμε διεθνείς επιχειρήσεις που είχαν στόχο την ε, σύλληψη κυβερνοεγκληματιών και βοηθήσαμε στο συντονισμό των ερευνών για πολύ μεγάλες και σημαντικές υποθέσεις κυβερνοεγκλήματος. Το κέντρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι κάτι στο οποίο θα σταθούμε αργότερα και το κέντρο που καλύπτει τις υπόλοιπες εγκληματικές δραστηριότητες όπως διακίνηση ναρκωτικών είναι ένα κέντρο που έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, βοηθούμε στην καταπολέμηση και του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γι' αυτό το έχουμε δημιουργήσει το Κέντρο Ηλεκτρονικού Οικονομικού και Χρηματοπιστωτικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της Ευρωπόλ. Να σας δώσω και μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων που στηρίξαμε. Τον Ιούνιο του 2019 έγινε μια πανευρωπαϊκή επιχείρηση κατά της διακίνησης ανθρώπων στην επικράτεια της Ένωσης. Η Ευρωπόλ είχε τον συντονιστικό ρόλο ε, της επιχείρησης εξάρθρωσης πύρας ε, που διακινούσε ανθρώπους με σκοπό την επαιτία. Είχαμε τη συνδρομή 15 κρατών μελών, τη συμμετοχή της Ισλανδίας και της Ελβετίας πέραν αυτών και ελέγξαμε 127.000 άτομα, πάνω από 600 οχήματα και πάνω από 100 τοποθεσίες. Το αποτελέσματα ε, είχαν να κάνουν με 34 συλλήψεις για διακίνηση και 36 συλλήψεις για άλλους λόγους. Εντοπίστηκαν επίσης 206 πιθανά θύματα εγκλημάτων, από τα οποία τα περισσότερα ήταν ανήλικα. Αυτά λοιπόν ε, ως ε, μία σύνοψη των δραστηριοτήτων μας. Επίσης, έχουμε συνδράμει στα κατημέλη σε θέματα που είχαν να κάνουν με την υγεία και με την ασφάλεια των τροφίμων. Διεξάγουμε λοιπόν έρευνες ε, μέσω ενός κέντρου το οποίο ειδικεύεται σε αυτό. Επίσης έχουμε ασχοληθεί και με θέματα πλαστογραφίας, ε, σε θέματα, ε, με θέματα παραποίησης φαρμάκων και τροφίμων. Βλέπουμε πως αυτό είναι μια τάση αρκετά ε, ανωδική. Επίσης, συνεργαστήκαμε με, την, με τις γαλλικές και φιλανδικές αρχές για εγκλήματα που είχαν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία και εδώ είχαμε επιτυχία πολλές συλλήψεις, εξάρθρωση αρκετών εγκληματικών ομάδων. Επίσης, σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, έχουμε παρατηρήσει μεγάλη κατάχρηση και παραβίαση των κανόνων και σε συνεργασία με τις υγειονομικέ αρχές των κρατών μελών καταφέραμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Άλλο ένα παράδειγμα της ε, δραστηριότητάς μας κατά της μαφίας, της Ντραγκέτα. Είχαμε την επιχείρηση Πολίνο το 2018, η οποία ήταν η μεγαλύτερη συντονισμένη δράση κατά μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Η επιχείρηση αυτή ήταν μοναδική, ήταν μια κοινή έρευνα από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές της κάτω χώρες, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο κατασχέσαμε περίπου 400 τόνους κοκαίνης και άλλων ναρκωτικών. Έγιναν αρκετές συλλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών της ε, μαφίας. Στην Ιταλία έγιναν 44 συλλήψεις και κατασχέθηκα ε, περιουσία 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπόλ επίσης δημιουργεί διασυνδέσεις. Έχουμε τους ε, υπεύθυνους διασύνδεσης, οι οποίοι βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ χωρών. Έχουμε την δυνατότητα να τους παρέχουμε στήριξη διμερώς και η υπηρεσία μας επίσης διαθέτει ένα εξωτερικό δίκτυο που βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίες Έχουμε περίπου 40 τέτοιες συμφωνίες και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται για άλλες 8 επιχειρηματικές ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επίση, για να στηριχτούν οι δραστηριότητέ μα, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Έχουμε λοιπόν ε, διάφορε ενημερωτικέ εκστρατείε στο διαδίκτυο για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο διαδίκτυο. Επίση, έχουμε ένα δίκτυο για την ε, καταπολέμηση ε, το περιπτώσεων απαγωγή για λίτρα. Είχαμε αρκετέ επιτυχίες και σε αυτόν τον τομέα από το 2016 μέχρι τώρα. Επίσης, η Ευρωπόλ κοιτάζει προς το μέλλον με μεγάλη φιλοδοξία. Τον Δεκέμβριο του 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική μας με μεγάλη πλειοψηφία διότι έχουμε καταφέρει να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες των κρατών μελών για μια πιο ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, για το καλό των πολιτών για την... και για να δώσουμε απαντήσεις και βοήθεια στα θύματα εγκλημάτων. Η Ευρωπόλ έχει πέντε στρατηγικούς στόχους και θα χρησιμοποιήσει στο έπακρο το κέντρο ε, πληροφοριών για ε, ποινικά ζητήματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα εστιάσουμε σε υποθέσεις προτεραιότητας στις πιο επικίνδυνες, στους πιο επικίνδυνους ε, εγκληματίες. Ε, νομίζω πως ε, με τις δυνατότητες που έχουμε κανένας εγκληματίας δεν θα μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Χρειάζεται όμως να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να αυξήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον χώρο της επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να δώσουμε το καλό παράδειγμα, καθώ επίση και να φροντίσουμε για τη χρηστή διακυβέρνηση εντό του οργανισμού μα. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα χρειαστεί ε, επαρκής χρηματοδότηση, επαρκής διαρκής χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν αυτό φαίνεται και στον προϋπολογισμό του οργανισμού μας για το 2020, όχι μόνο της Ευρωπόλ αλλά και των συνεργαζόμενων με εκείνη οργανισμών. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνει ξανά η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας ε, εν ώψη του νέου προϋπολογισμού. Επίσης, έχουμε εννέα οργανισμούς, Frontex, Euliza, Θεμελιώδη Δικαιώματα, CIPOL, CVDA, AG, Eurojust, EASO και εμείς, η Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ έχει την προεδρία φέτος αυτού του δικτύου και έχει εντοπίσει ορισμένους κεντρικούς τομείς στους οποίους θέλει να δώσει έμφαση. Διαλειτουργικά συστήματα πληροφορική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, διότι θέλουμε να παρέχουμε μια καλή στρατηγική για το πώς μπορούν να συνεργαστούν προ όφελο των πολιτών οι εννέα αυτοί οργανισμοί. Θα σας παρουσιάσουμε το έγγραφο στρατηγικής πολύ σύντομα στις αρχές του επόμενου έτους. Επίσης, συζητούμε και θέματα ad hoc, όπω του τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ε, στους διάφορους ε, οργανισμούς, πώς μπορούμε να φέρουμε την καινοτομία στα, στους διάφορους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συζητούμε θέματα πολυμορφίας, που είναι πολύ σημαντικά. Μετά, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλου με τους άλλους ε, οργανισμούς επιβολής του νόμου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη Frontex. Με τη Frontex μάλιστα έχουμε και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Με την ΕΑΣΟ έχουμε, κάνουμε από κοινού εκθέσεις αναλυτικές. Υπάρχει συνεργασία με τη Eurojust για δικαστικά και αστυνομικά ζητήματα. Με τη ΣΕΠΟΛ επίσης ε, διοργανώνουμε από κοινού οικοδόμηση ικανοτήτων. Με την ε, εκτίμηση επίσης από κοινού την, της κατάστασης σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών. Και συζητούμε με την ΕΠΟ για τη νέα της κατεύθυνση. Τώρα, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Μας βοηθάει, για παράδειγμα, σε θέματα κατάρτισης ε, των ε, υπαλλήλων που μεταβαίνουν στα hotspot. Η Ευρωπόλη έχει μία έκθεση εμβληματική σχετικά με την κατάσταση στην, δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο του 2017 ξεκίνησε να δημοσιεύεται για πρώτη φορά και πέρυσι είχαμε ε, την ε, επόμενη. Το 2019 έχουμε δει μία κάποια εμφάνιση μια κάποια μείωση του συνόλου των ε, τζιχαδιστικών ε, τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά μια αύξηση των ακροδεξιών ε, τρομοκρατικών επιθέσεων. Βέβαια τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ποτέ. Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία γι' αυτό. Έχει μειωθεί ο συνολικός αριθμός επιθέσεων, όμως ο αριθμός των επιθέσεων που είχαν σχεδιαστεί αλλά καταφέραμε να αναχαιτήσουμε έχει αυξηθεί. Επίσης, επιθέσεις με χημικά δείχνουν πως ορισμένες μεμονωμένες τρομοκρατικές ομάδες επιμένουν να απειλούν τις ε, ζωές των πολιτών. Επίσης ε, υπάρχουν επιθέσεις από πνευματικά ασταθείς ανθρώπους οι οποίοι αντιγράφουν τζιχαντιστικές επιθέσεις βλέπουμε ότι τα όρια μεταξύ διαδικτύου και ε, μη αρχίζουν και θολώνουν και κάνουν πολύ πιο δύσκολο το έργο μας. Υπάρχουν άτομα τα οποία επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου, όμως είναι οργανωμένα σε offline ομάδες ε, οι οποίες έχουν περάσει από στρατιωτική εκπαίδευση για τρομοκρατικές πράξεις στις εμπόλεμες ζώνες του Ιράν και της Συρίας παιδιά, ανήλικοι, είναι εκτεθειμένα σε τζιχαντιστική ιδεολογία, σε τρομοκρατική ιδεολογία και ενδεχομένως ε, αποτελέσουν απειλή για το μέλλον. Έπειτα έχουμε και την ε, καταπολέμηση του ακροδεξιού εξτρεμισμού, βίαιου εξτρεμισμού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει σχετικά χαμηλός αριθμός επιθέσεων, όμως βλέπουμε αυξητικές τάσεις τα τελευταία τρία χρόνια. η ακροδεξιά δραστηριότητα δεν έχει δείξει τόσο αιματηρές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά ε, πλήση εγκεφάλου, αλλαγή νοοτροπίας ε, και μέσω της ρητορική μίσους που κατευθύνεται σε ε, Προσπαθούμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε όλα αυτά και να προστατεύσουμε τα θύματα, ιδιαίτερα του τζιχαντισμού. Θα σταματήσω την παρέμβασή μου εδώ. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, θα χαρώ πολύ να ακούσω σχόλια και συμβουλές για το τι μπορούμε να κάνουμε στην υπηρεσία μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεμπόλ για την προσπάθειά σας αυτή να συγκρατηθείτε και να τηρήσετε και το χρόνο σας. Ο χρόνος που πιέζει γενικώ στην Επιτροπή μας. Θυμίζω ότι έχουμε κατάλογο μιλητών και μακρύ right after the first round of... Ο πρώτος γύρος πάντα είναι οι ε, συντονιστές και μετά απαντήσεις. Παρακαλώ και τους συντονιστές λοιπόν να χωρέσουν σε 1,5 λεπτό την ερώτησή τους και ο επόμενος γύρος ένα λεπτό για τον καθένα, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Including the following point of the order of the day. So we get Προχωρούμε λοιπόν. Συντονιστές. Η κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, όπως μόλις ακούσαμε, ξέρουμε όλοι ότι οι απειλές στην εσωτερική ασφάλεια παραμένουν πολύ ψηλέ. Ε, στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο εργαστήκαμε για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, ας πούμε με την αναθεώρηση ε, της ε, ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής και αυξήσαμε τους πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους στο Frontex και επομένουν να γίνουν κι άλλα. Ωστόσο, δεν είδαμε το ίδιο για την εσωτερική ασφάλεια σε ανθρωπίνους πόρους και οικονομικούς. Και η Ευρωπόλ είναι πραγματικά ε, παράδειγμα χαρακτηριστικό. Ε, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε γενναία χρηματοδότηση, επένδυση στην Ευρωπόλ για να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία για την επιβολή του νόμου, για την καταπολέμηση του ε, λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του ξεπλήματος χρήματος, της ε, τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αναφερθήκατε στον προϋπολογισμό που προτείνεται για το 2020 και ε, το αίτημα να μειωθούν σημαντικά οι συμβασιούχοι στην Ευρωπόλ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό τι σημαίνει και τι επίπτωση θα έχει στη λειτουργία του οργανισμού σας αυτό και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε να καταφέρουμε να συγκεράσουμε τέτοιες προτάσεις δημοσιονομικές με τις ανάγκες της όλο αυξανόμενες. Για την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών αναφερθήκατε στο τέλος αυτό. Μας δώσατε μερικά παραδείγματα για τη συνεργασία με την ηγεσία της Europol, με άλλους οργανισμούς εσωτερικών και δικαιοσύνης. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο για το μέλλον Ακούμε όλο και περισσότερο, ε, ιδιαίτερα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αν μπορούν κάποιες γραμμές από τον προπολογισμό να αναδιαταχθούν για να βοηθήσουν ε, έτσι εμπροστοβαρός κάποιους οργανισμούς που χρειάζονται χρήματα στην αρχή της θητείας τους και λιγότερο στο τέλος. Έχετε εσείς τέτοια ζητήματα ή είναι όλα εντάξει, η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξεκινήσω με ένα μικρό σχόλιο σε ό,τι αφορά το, τη χρηματοδότηση της Europol. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, πολύ αμφιβάλλω για την αποτελεσματικότητα της ε, διαρκούς αύξησης της χρηματοδότησης της Europol. Φυσικά καταλαβαίνω ότι οι εθνικές αρχές και η αστυνομία και το δικαστικό σώμα δεν έχουν στη διάθεσή τους τους πόρους που χρειάζονται. Άρα, αναρωτιέμαι πώς μπορούμε αυτό να το διαμορφώσουμε ε, με αποτελεσματικό τρόπο για την εργασία επιτόπου. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί έχουμε πολλά καινούργια μέλη. Είπατε και μιλήσατε για την υποστήριξή σας προς τη Μάλτα, τη Σλοβακία, σε ό,τι αφορά τους ε, δημοσιογράφους που δολοφονήθηκαν. Πείτε μας συγκεκριμένα πώς υποστηρίζετε τις χώρες αυτές. Πού βρισκόμαστε επίσης και στις ε, έρευνες που γίνονται για τα θέματα αυτά. Έχουμε βρει τελικά ποιοι είναι οι πέτοι οι, ποιοι κρύβονται και ποιοι είναι αυτοί που έδωσαν εντολή για τι δολοφονίε αυτές. Αναφέρεται επίσης στην ε, παράνομη διακίνηση ανθρώπων και σε ό,τι αφορά επίσης ε, τους ε, ανηλίκους, τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, πώς υποστηρίζεται τα άτομα αυτά και τους ανηλίκους αυτούς. Επίσης βλέπουμε μεγάλη ροή ε, ενηλίκων που έρχονται παράνομα. Από τη μία ο κόσμος ε, παραπονιέται για τους παράνομους μετανάστες, από την άλλη βρίσκουν τις εργασίες στην κοινωνία μας. Ε, θα ερευνήσετε λοιπόν τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εντφέλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. σας ευχαριστώ, κυρία Ντεμπόλη, που βρίσκεστε εδώ. Τρεις ερωτήσεις σύντομες έχω να κάνω αναφέρθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές σε ό,τι αφορά τις έρευνες για τη τηλεφωνία ε, στην ε, Μάλτα και στη Σλοβακία. Στη Μάλτα, όλους ιδιαίτερους, πείτε μας. Η Europol εξακολουθεί να συμμετέχει στις έρευνες. Ε, έχετε την αίσθηση ότι είστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή σας, την πρόσβαση στις πληροφορίες και σε όλα τα τμήματα της έρευνας. Κατά δεύτερον, οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα προσωπικά και η διάδοση αυτών είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Βλέπουμε ότι διαρκώς ανακύπτουν θέματα για την ακρίβεια και την εμπιστευτισμότητα των ε, στοιχείων των δεδομένων αυτών και στη δανεική περίπτωση της Δανίας ε, και στην περίπτωση της Γερμανίας ε, αλλά και σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των αρχών. Ξέρουμε ότι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με το Πολωνικό Δικαστικό Σώμα, για παράδειγμα. Όλα αυτά πώς επηρεάζουν τη δική σας δουλειά. Γιατί η Κομισιόν λέει ότι υπάρχει η ότι θεωρητικά υπάρχει συμμόρφωση, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά, ξέρουμε. Κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι κυνηγάται εγκληματία και παρόλα αυτά εξακολουθούνται να έχετε τα συστήματα χρυσών ε, θεωρήσεων και χρυσών ε, διαβατηρίων που ανοίγουν με την πίσω πόρτα την ε, πρόσβαση στους εγκληματίε και μεγάλο εγκληματίε μάλιστα. Άρα αυτά τα χρυσά διαβατήρια αυτές οι χρυσές θεωρήσεις πώς θα αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μελητρία. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ντεμπόλα για την παρουσίαση τη και εγώ έχω κάποιε ερωτήσει να κάνω. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σκέλο τη εξωτερική συνεργασία. Ε. Ο κόσμο ε, βγαίνει στο εξωτερικό όλο και πιο πολύ. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά τα οποία φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τυχάνουν κατάχρηση για άλλους σκοπούς και πολιτικούς σκοπούς. Αυτό πώς θα επιληθεί στους κόλπους της Europol και αυτό μιας και η Europol συνεργάζεται όλο και πιο πολύ με την Frontex και την EASO. Εδώ υπάρχουν ε, μεγάλοι όγκοι δεδομένων που ανταλλάσσονται και ενδεχομένως να είναι σε κίνδυνο ή την τεσάσυλο ή μετανάστευση μετανάστες, πρόσφυγες σε ό,τι αφορά και τις χώρες προέλευσης. Άρα η Europol ε, συμμορφώνεται με τον σχετικό χάρτη και τον ε, κανόνες για την ευρωπαϊκή ιδιωτική σφαίρα σε ό,τι Εδώ Europol είναι να ξαναθέσουμε τις προτεραιότητές μας γιατί θα πρέπει να κάνουμε αυτή την άσκηση για την, τον ορισμό των προτεραιότητων μας με τα κρατη Θα πρέπει οι πελάτες μας να αποφασίσουν ποιες ε, επενδύσεις δεν θα γίνουν πλέον στο IT, στην κινητομία, σε ό,τι αφορά ε, την ανάπτυξη των ε, γραφείων στο hotspot, υποστήριξη των κρατών μελών με ε, στρατηγικές συναντήσεις, αποστολές, ε, κόστος των αποστολών, ε, διαχειριστικό κόστος, λύσεις ενίσχυση της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Αυτό φυσικά θα σημαίνει επιπλέον υπαλλήλου, το οποίο δεν γίνεται με λιγότερο προϋπολογισμό. Και επίσης θέλουμε στόχους υψηλόβαθμους και εδώ χρειαζόμαστε πιο πολύ χρηματοδότηση το πρόγραμμα πέρσι, για παράδειγμα, είναι η συνέχιση του προγράμματος Ήρμα που έχουμε για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει φυσικά. Δεύτερη ερώτηση για την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών με τη Frontex. Έχουμε πολύ καλό σχέδιο δράσης που ορίζει τους διάφορους τομείς κλειδί για τη συνεργασία, καινοτομία, στρατηγική ανάλυση, συνεργασία και εξωτερικές σχέσεις. Συχνά συνεργαζόμαστε με τη Frontex σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες αντικτύπου. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Frontex και της Europol. Η Europol λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει ο κόμβος ποινικών πληροφοριών για τις αστυνομικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Frontex είναι τα μάτια για τα αυτιά της κοινότητας επιβολής δικαίου στα σύνορα με την ΕΑΖΟ. Έχουμε κάνει κοινέ εκθέσεις ανάλυσης σε ό,τι αφορά θέματα πολύ σημαντικά. Και επίσης προωθήσαμε και τα θέματα αυτά με τις συνδεδεμένες χώρες με την Ευρώπη του Σέγγιν. Επίσης έχουμε από τη Eurojust τα δικαστές ε, στην υπηρεσία μας ε, για θέματα κυβερνοεγκλήματος και επίσης ε, συνεργαζόμαστε μαζί τους ότι αφορά το κυβερνοέγκλημα και τις εγκληματικές δραστηριότητες. Με τη ΣΥΠΟΛ επίσης έχουμε συνεργασία, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι η ΣΥΠΟΛ έχει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά θέματα εκπαίδευση. Εμεί δίνουμε εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την υπηρεσία για τα ναρκωτικά, που μα αναφέρει τι γίνεται με τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε μια κοινή έκθεση. Και με τον δημόσιο εισαγγελέα θα θέλαμε να ξέρουμε σε τι βαθμό θα πρέπει να υποβάλουμε τις αναλυτικές εκθέσεις που αναφέρονται στον κανονισμό. Όταν θα ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα, θα υπάρχει συνεργασία με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Επίση, με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχουμε στρατηγική συνεργασία, έχουμε τι συστάσει τη υπηρεσία, τι οποίε και τι ε, επιβάλλουμε και έχουμε και συνδέσμους ε, στα διάφορα hotspots. Θέλουμε να αποφύγουμε πάντα ε, αλληλεπικάλυψη καθηκόντων με τις υπηρεσίε αυτές. Συνεργαζόμαστε όλο και πιο στενά σε ό,τι αφορά για την γενοτομία. Έχουμε στην συνεργασία με τη Frontex, με το Ιουλίζα και με τα κρατημέλη. Και ορίζουμε ποιος τελικά καθορίζει τι γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν από τη Europol να αποτελεί την πλατφόρμα για την αστυνομική συνεργασία. Άρα εξετάζουμε από τα κράτη-μέλη ποιος είναι ειδικό σε τι και προσπαθούμε να καινοτομήσουμε σε διάφορους τομείς. Προκειμένου οι καινοτόμες λύσεις να είναι στη διάθεση των διαφόρων αρχών και υπηρεσιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μάλτα και τη Σλοβακία, η Γεροπόλου. Μας ζητήθηκε να υποστηρίξουμε τις ε, έρευνες επιτόπου και στη Μάλτα και στη Σλοβακία. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποια είναι η δική μας θέση, ποια είναι η δική μας εντολή, αν θέλετε. Δεν έχουμε ε, εντολή επιβολής. Αυτό είναι στα χέρια της εθνικής ε, αρχής. Εμείς, σε πρώτη φάση, μόνο όταν μας ζητείτε μπορούμε να παρεμβούμε. Καταρτήσαμε λοιπόν ένα σχέδιο δράσης με τους ερευνητές, κάναμε αναλυτικό έργο, συντονισμό των, ε, της συλλογής στοιχείων, διευκόλυνση και επιβεβαίωση των στοιχείων. Άρα πιο πολλά είναι αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και σε ό,τι αφορά την ε, δικαιοσύνη και την αστυνομία, για παράδειγμα, κρυφές αποστολές, επιβολή μέτρων, Υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις θέματα τα οποία συνδέονται με τη γλώσσα. Δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε πότε θα γίνουν οι ε, επιχειρήσεις. Εμείς μόνο προτάσεις μπορούμε να κάνουμε. Κάναμε σημαντικές προτάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή ε, στοιχείων και την ανάλυση στοιχείων. Και η συνεργασία μας θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική. Είναι σε εξέλιξη ακόμα. Είμαστε στη διάθεση της κοινότητας επιβολής ε, του νόμου. Δεν μπορούμε όμως εμείς να αποφασίζουμε τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των ερευνών. Αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Προστασία των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μας ελέγχουν ε, διάφορες ε, μηχανισμοί. Έχουμε τον DPO μας, ε, τον, μηχανισμό τον άτομο που είναι υπεύθυνο για την συντονισμό των στοιχείων αυτών. Επίση, υπάρχει η κοινότητα προστασία των δεδομένων, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία Δεδομένων και υπάρχει και την ενότητα τα άτομα να υποβάλουν ερωτήματα προς την υπηρεσία μας και εμείς στη συνέχεια εξετάζουμε κατά πόσον μπορούμε να δώσουμε μια σωστή απάντηση στα άτομα αυτά. Η προστασία των δεδομένων είναι πολύ υψηλού επίπεδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα πολύ δυνατό σύστημα το οποίο ορίζει ο κανονισμός. Κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να τηρήσουμε της στάσεις του EPPS και επίσης ε, προκειμένου ο αξιωματούχος για θέματα προστασίας δεδομένων να είναι δίπλα μας για να μπορεί να αξιολογεί πώς γίνεται η διαχείριση των δεδομένων. Έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες. Υπάρχει και το θέμα της ε, οικονομικής επένδυσης ε, που χρειάζεται στον τομέα αυτό προκειμένου να τηρούνται ενήμερα όλα αυτά τα συστήματα. Το ερώτημα για το PNR τώρα. Έχουμε τη γραμματεία του ατυπού δικτύου για το PNR για την ανάπτυξη του συστήματος στις διάφορες χώρες. Ε, θέλουμε να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τα συστήματα τα δικά τους για την τρομοκρατία και την ανταλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία αριστερής, αριστερού, αριστερών και δεξιών εμείς ε, εξαρτώμαστε από τι πληροφορίε που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Όταν μιλάμε για σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, η Europol μπορεί να παρέμβει μόνο όταν υπάρχει εμπλοκή δύο κρατών μελών. Όταν ε, ε, μιλάμε για τρομοκρατία, χρειάζεται η εμπλοκή ενό κράτου μέλου. Είναι απαραίτητο λοιπόν από κοινού το κράτο μέλο να εξετάσουμε τι είδου ενέργεια χρειάζεται, τι είδου επιχείρηση χρειάζεται για την εντοπίση του κλίματος. Το θέμα των μεταναστών, τη διακίνηση, ε, είναι τεράστιο θέμα για μα. Κάνουμε λοιπόν μεγάλε προσπάθειε με το κέντρο για τη διακίνηση ανθρώπων και προσπαθούμε να βρούμε του διακινητέ πίσω από του μετανάστε και του πρόσφυγε. Έχουμε μια κοινή ομάδα σύνδεση ε, για τα θέματα αυτά, προκειμένου οι χώρε οι οποίε πλήττονται ιδιαίτερω να μπορούν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και να συζητούν τα θέματα που ανακύπτουν και ελπίζω έτσι να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε ε, κύριε Αντεμπόλ που σέβεστε το χρόνο και ελπίζουμε να σας μυθούν ε, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Τουλάχιστον 13 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ένα λεπτό έκαστος για να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Παρακαλώ να περιορίσετε τη διατύπωση την ίδια της ερώτησής σας να χωράει σε ένα λεπτό. Η κυρία Παγάσα Ορτούντου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και συγχαρητήρια για την έκθεση. Είναι σαφέστατη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η έκθεση. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας. Ε, πολύ σαφίστηκε και στις απαντήσεις ήσασταν. Έχω να ρωτήσω για το ρόλο της Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά την αναζήτηση πληροφοριών επιτόπου ε, στο Ιράκ και τη Συρία. Πώς θα συντονίζετε αυτά, γιατί χιλιάδες Ευρωπαίοι εκεί έχουν γίνει τρομοκράτες. Και από τη στιγμή που κατέρευσε το Ισλαμικό Χαλιφάτο, κινδυνεύουν να μείνουν ατιμόρυτες πολλές εγκληματικές ενέργειες, σοβαρότατες παραβιάσεις εκεί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Μωράε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ντεμπόλε για το έργο της γενικότερα και την ομάδα της, ε, το επιτελείο στη Europol. Το εκτιμούμε βαθύτατα. Απαντώντα στην κυρία Μετσόλα για τον προπολογισμό, είπατε κάτι και θέλω να επανέλθω κυρίω για του νέου βουλευτέ. Ε, γιατί το JPSG, ε, η δομή που έχουμε φτιάξει, ε, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τον προπολογισμό του 2020. Εσείς είστε σε μια πολύ δυσχερή θέση. Θα πρέπει να λέτε ότι χρειάζεστε περισσότερα χρήματα και το αναλύετε αυτό λεπτομερώς. Έλα, να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν ισχύει ότι η Ευρωπόλ ε, έχει πολύ ψηλό προφίλ, ε, είναι μοναδικός οργανισμός, δεν έχει δυνατότητα επιβολής. Ε, συλλογή πληροφοριών είναι το έργο της, είναι σχετικά μικρή και θα πρέπει να καταλάβουν και τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου πόσο μικρή οργάνωση είστε. τα κράτη-μέλη κάθε τόσο ζητούν πολλά περισσότερα από τη Europol, όχι μόνο για τα hot spots, αλλά επιβαρύνουν πολύ τον προπολογισμό τη. Μήπω υπάρχει μια δυσαναλογία εδώ ε, στην επιβάρυνση και μπορείτε να μα εξηγήσετε τι είναι αυτό και πώ μπορούμε και γιατί να σας βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Εκτελεστική Διευθύντρια για την παρουσίασή σας. Θα συνεχίσω στα ρουμανικά, στη μητρική μου γλώσσα. Sorry, the mic. Yes. Conform datelor... Έλεγα, λοιπόν, ε, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει η κυρία Στρογκάρου, πέρσι πάνω από 20.000 άνθρωποι είναι θύματα του τράφικη στην Ευρώπη. Το 68% είναι γυναίκες και νεαρά κορίτσια. Με πρώτη θέση τη Ρουμανία ως χώρα προέλευσης, στη συνέχεια ε, Πολωνία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και κάτω χώρες. Έχω την εξή ερώτηση λοιπόν. Ε, αναλύοντας αυτούς τους αριθμούς διαπιστώνουμε ότι χωρίς χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχουν τεράστια προβλήματα. Τι στρατηγική έχει η Ευρωπόλ για το ερχόμενο διάστημα έτσι ώστε να καταπολεμήσει άμεσα και αποτελεσματικά αυτή τη διακίνηση ανθρώπων, το trafficking. Δεύτερον, η τεχνολογία 5G στα κινητά τηλέφωνα. Ποια είναι ε, τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα, ποιες είναι ευάλωτες στις και πώς προετοιμάζεται η Europol και τι ε, πόρους χρειάζεται για να προετοιμαστεί στις νέες τεχνολογίες. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος ε, Μπράιερ. Για το ίντερνετ έχετε μια μονάδα εκεί. Όταν βρίσκεται ένα ηλεκτρονικό έγκλημα, αυτά τα λέτε και στην αστυνομία και το δεύτερο αφορά ε, την κράτηση, διατήρηση δεδομένων. Έχετε μια περιορισμένη διατήρηση δεδομένων, έτσι το ονομάζετε Και εξαιρείται κάποιους επαγγελματίες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξεκάθαρα είπε ότι ε, παραβιάζεται έτσι ε, τα δικαιώματα ε, των ε, ανθρώπων που ούτε κατά διάνοια, ούτε μακράν δεν συνδέονται ε, με οργανωμένο έγκλημα. Γιατί το κάνετε αυτό και τι θα γίνει. Δέχεστε αυτή την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη Europol και πού βασίζετε τη δράση σας επ' αυτού, σε ποια νομικά ερίσματα. Ευχαριστώ. Από την Γκουε, η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Διευθύντρια, θέλω να ρωτήσω το ρόλο της Ευρωπόλ ως διαχειριστή πολύ ευαίσθητων δεδομένων και τι σχέση έχετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων, EDPS. Είδαμε πέρσι κάποιες έρευνες και με τα δικά σας συστήματα προφοριών, που δεν έχετε μόνο υπόπτους και καταδικαστέντες αλλά πιθανούς μελλοντικούς εγκληματίες. Ποιοι είναι αυτοί, πώς ορίζονται και ποια είναι τα εχέγγυα που έχετε για να ε, αποφύγετε profiling σε σχέση με την εθνοτική προέλευση. Και επίση τι γίνεται με το πρόγραμμα επιχειρησιακής ανάλυσης για τους επιβάτες και τους ταξιδιώτες. Τους ξένους μαχητές και τους τρομοκράτες πώς τους αναγνωρίζετε και ποιες είναι οι εγγύσεις. Και αυτό το τελευταίο που ακούσαμε από το φίλο ε, του ID για την αριστερή τρομοκρατία, την ακροαριστερή, μάλλον δεν διάβασε την έκθεση. Εσείς τι λέτε για τις εθνικές κυβερνήσεις. Γιατί λέτε για μια βίαιη ε, ε, αποσχιστική δραστηριότητα στην Ισπανία. Αυτά ποιος σας τα έχει δώσει, ο κύριος Λέναρτς. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου ερώτηση έχει να κάνει με το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Έχω διαβάσει στο πρόγραμμα της Ευρωπόλου ότι θέλετε να ε, τροποποιήσετε την πρόσβαση στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιούμε καλά. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε το σύστημα και πότε μπορούμε να περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έπειτα, το επικαιροποιήσαμε το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν πέρυσι. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει δώσει καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρωπόλ. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την διαδικασία αυτή και τι νέε δυνατότητε που θα έχει το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Πού βρίσκεστε, τι, ε, πόσο απέχετε μέχρι να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε στο 100% όλε τις δυνατότητές του. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανίτσι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντεμπόλ, για την παρουσίασή σας σχετικά με τι δραστηριότητε τη Ευρωπόλη. Εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Τώρα σε ό,τι αφορά την πρόσφατη συμμετοχή σας στην Σύνοδο με τι αρχέ των ΗΠΑ όπου συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και πρόσβαση στην πληροφορία ε, καθώς και το ίντερνετ των πραγμάτων και το δίκτυο 5G. Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα έτσι ώστε να διασφαλίζετε η ασφάλεια αυτών των ε, τεχνολογιών, αυτών των συσκευών για να μην πέσουν στα χέρια τρομοκρατών. Μας είπατε επίσης ότι έχετε διοργανώσει διάφορες επιχειρήσεις όπου έχουν εξουδετερωθεί εγκληματικές ομάδες, έχουν αποτραπεί επιθέσεις. Εσείς θεωρείτε πως στο μέλλον θα υπάρξουν περισσότερες ε, τέτοιες οργανωμένες επιθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντεμπόλ, θα μιλήσω ε, Ολλανδικά ω ε, Βελγίδα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχετε τη θέση αυτή και για την εργασία που κάνετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πολλέ ερωτήσει ακούσαμε για τη χρηματοδότηση, γιατί για μένα το θέμα αυτό αφορά και την ιστορική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αλλά ένα έντεκο, ενδέκατο δίνουμε σε σχέση με αυτά που δίνουμε για την ιστορική ασφάλεια. Και μα αναφέρετε μία σειρά εργασιών που δεν θα μπορείτε να κάνετε πλέον, γιατί δεν πήρατε την χρηματοδότηση που θέλετε. Με ανησυχεί αυτό. Δηλαδή, τελικά τι, το IT και η Κοινοτομία θα τα διαγράψουμε, κατά πολέμηση των ναρκωτικών δεν θα μπορέσουμε να τα συνεχίσουμε. Η ενημέρωση βασικών προγραμμάτων δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Μπορείτε να μα εγγυηθείτε ότι η Europol αυτή τη στιγμή με τη χρηματοδότηση που έχει λάβει θα μπορέσει να φροντίσει την ιστορική Ένα ασφάλεια γιατί ιδάλω θα πρέπει να αναλάβουμε κατεπηγόντω δράση. Ένα άλλο θέμα. Ξεκινάει η νέα θετία και η Europol ε, παίρνει όλο και πιο πολλές επιπρόσθετες εντολές. Μπορείτε λοιπόν να επιτελέσετε όλα αυτά τα καθήκοντα γιατί εμείς θέλουμε να φροντίσουμε ότι θα είστε στη θέση να κάνετε τις εργασίες σας. Θέλουμε λοιπόν να προσαρμοστεί η εντολή σας αυτή για να μπορέσετε να την επιτελέσετε, να την εκτελέσετε. Κατά τρίτον, 10.000 αγνοούμενα παιδιά προσφύγων. Θα ήθελα να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πίτερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ Βέλγο είμαι, αλλά θα μιλήσω αγγλικά τώρα. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το δίκτυο 5G. Είμαστε όλοι θετικοί στην εισαγωγή του 5G, υπάρχουν όμως πολλά αλλά, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι προκλήσεις βλέπει στο πλαίσιο της εισαγωγή του 5G και πώς η Ευρωπόλ θεωρεί ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Μετά, έχω και μία ερώτηση για τις δευτερογενείς ε, μεταναστευτικές ροές. Έχουμε παρατηρήσει αύξηση αυτών των ροών τελευταία. Η Ευρωπόλ λοιπόν θεωρεί πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια ως αποτέλεσμα αυτών των δευτερογενών μεταναστευτικών ροών. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα και μετακινούνται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς, λοιπόν ε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, πώς μπορούμε να αγγίθουμε την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χούκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να εστιάσω στην απάτη και να ρωτήσω για τη σχέση τη Ευρωπόλη με τις τράπεζες. Έχουμε πολλά περιστατικά απάτης, μικροαπάτης ε, για μερικές χιλιάδες ε, λίρε που σημειώνονται διασυνοριακά. Ο αριθμός των ε, συλλήψεων είναι Μικρό. Πολλές φορές ε, βέβαια όταν γίνονται κάποιε συλλήψει, μπορούμε να παρακολουθήσουμε το τι έχει γίνει, από ποια τράπεζα έχει ξεκινήσει, ποια τράπεζα έχει πάει, ομω οι τράπεζε δεν θέλουν να δώσουν στοιχεία. Η Ευρωπόλη πώ μπορεί να τι ενθαρρύνει να το κάνουν. Έπειτα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Θέλω να ρωτήσω, μα ε, είπατε μάλλον ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα θύματα. Όμω η αντιμετώπιση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξέσπασε πρόσφατα ένα σκάνδαλο για τα θύματα απάτη, τα οποία όχι μόνο έπεσαν θύματα απάτης, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε με τις υποθέσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν τι ε, νομίζετε πώς πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Ε, κυρία Κελέρ, ευχαριστώ. Μετά ε, τους Σίπελ, Μωράες και Βότμαν, θέλω και εγώ να αναφερθώ στον προϋπολογισμό σας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 20% κάτω του δικού σας σχεδίου προϋπολογισμού. Εσείς λαμβάνατε υπόψη τις σημαντικές σας ανάγκες, και ε, οι πολλές ερωτήσεις των συναδέλφων δείχνουν ότι αντιμετωπίζετε τεράστιες προκλήσεις και ποιες είναι αυτές. Η προστασία, η διαχείριση των δεδομένων, ο συντονισμός, η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών αλλά και με τρίτες χώρες. Οπότε, κυρία Γενική Διευθύντρια, πώς μπορείτε να εξηγήσετε αυτή την απόσταση ε, ανάμεσα στις αποστολές σας που αυξάνονται και τα χρήματα. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί σε αυτή την ψελίδα. Κύριε κύριος σαν τελευταίο λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Ντεμπόλε για την εισαγωγή. Η πληροφορία και ανταλλαγή δεδομένων είναι κλειδί απολύτω όπως το είπατε και εσείς στα σχόλιά σας. Αλλά βλέπουμε και πολλά παραδείγματα όπου τα κράτη-μέλη δεν μοιράζονται τις απαραίτητες προφορίες για να καταπολεμήσουν, να προλάβουν ένα οργανωμένο έγκλημα, ακόμα και μια τρομοκρατική ενέργεια. Πώς θα βεβαιωθείτε ότι τα κράτη-μέλη μοιράζονται τις προφορίες που υποτίθεται ότι πρέπει να διαβιβάζουν. Ε, νομίζω ότι έχετε την απαραίτητη εντολή για να το εξασφαλίσετε αυτό. Και δεύτερο και πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Ε, οι βάσεις δεδομένων ε, σε κινητές συσκευές. Ε, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση από τα κράτη-μέλη εσείς τι θα κάνετε και πώς προβλέπετε εκεί να έχουν Σε Ευχαριστώ πολύ. Επανερχόμαστε στην εκτελεστική διευθύντρια. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων αν μας βοηθήσετε και μέσα σε ένα δεκάλεπτο αποφαντήσετε για να έχουμε και λίγο χρόνο για το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που μας απομένει για σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά τα χρηματοδότηση και για να απαντήσω και στην ερώτηση του κ. Μωράης. Ο αριθμός των προσωρινών υπαλλήλων είναι 546. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι συμβασιούχοι υπαλλήλοι εργάζονται με τα καθημερινά θέματα στο τρία κέντρα. Το Κέντρο κυριμερνό εγκλήματος, το Διακίνησης και στο IOU. Και οι προσωρινοί αυτοί οι υπάλληλοι είναι μαζί μας για εννέα έτη. Είναι από τον κλάδο της επιβολής του νόμου, είναι αστυνομικοί, έχουν αστυνομικό υπόβαθρο. Έχουμε επίσης συμβασιούχους που είναι στην υποστηρίξη κυρίως. Αυτοί οι συμβασιούχοι τους έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 208 τέτοιους συμβασιούχους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να τους περιορίσουμε σε 148. Αυτό είναι τεράστιο θέμα για μας, γιατί αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που μας υποστηρίζουν από πλευράς ε, IT για την ανάπτυξη επίσης ε, των συστημάτων, επίσης ε, ε, διοργανώνουν τις αποστολές, διοργανώνουν τις συναντήσεις μας, τις στρατηγικές συναντήσεις, τις διαχειριστικές συναντήσεις. Ύστερα έχουμε τους εθνικούς αποσπασμένους, οι οποίοι πληρώνονται από τα κρατημέλη και εμείς πληρώνουμε μια διατροφή και τη στέγασή τους. 117 έχουμε τέτοιους. Ύστερα έχουμε 178-179 ε, αξιωματικούς συνδέσμους από τρίτες χώρες, οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου ανεξάρτητοι, έχουν ε, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις, ε, τα δικτυά μας, στο ΣΧΕΝΑ, τα εργαλεία της Europol, έχουν πρόσβαση στα κεντρικά μας και μπορούν να συνεργάζονται διμερώς έχουν επίσης ε, στη διάθεσή τους ε, τις εγκαταστάσεις ε, της Europol 190 και έχουμε περίπου 30-40 άτομα εσωτερικούς ασκούμενους από πανεπιστήμια, πανεπιστήμια που έρχονται να εκπαιδευτούν σε θέματα Europol. 80% των θέσεων είναι σε θέσεις υποστηρίξης σε θέματα δικαίου δηλαδή και γενικά λαμβάνουμε καλά σχόλια από τους ελεγκτές ευρωπαϊκού επίπεδου σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της μείωσης της χρηματοδότησης. Θα είναι μεγάλος για την υπηρεσία γιατί έχουμε όλο και πιο μεγάλα όλο και πιο πολλέ εθνικέ αρχέ ε, από τα εθνικά τελωνία, από την εθνική αστυνομίες που μα ζητούν να επέμβουμε. Γιατί είναι πεπισμένοι ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία και φυσικά θέλουμε να, να βρίσκουμε και καινοτόμε λύσει από κοινού. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ζήτηση και φυσικά όταν θα μειωθεί ο προπολογισμό, αυτό θα έχει αντίκτυπο για δηλαδή το τι μπορούμε να κάνουμε σε λειτουργικό επίπεδο. Ήδη το βλέπουμε αυτό online. Καλούμαστε καθημερινά να αποφασίσουμε ποιο ποτέ θα, θα σώσουμε. Τέτοιες ε, επιλογές κάνουμε σε καθημερινή βάση. Σε άλλο επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις ε, οργανωμένες ομάδες εγκλήματος, ε, έχουμε ένα σύστημα προτεραιοτήτων όπου μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις περιπτώσεις άνω της προτεραιότητας. Δεν έχουμε δυνάμεις για παραπάνω σε ό,τι αφορά το EDPS και την προστασία των δεδομένων στην υπηρεσία μα. Έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για δικλείδε ασφαλεία για την προστασία των δεδομένων στον κανονισμό τη Europol. Για εμά, λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά να τα παρακολουθούμε καθημερινά. Έχουμε τον αξιωματούχο για την προστασία των δεδομένων μέσα στο γραφείο, ο οποίος καθημερινά εκτιμά το πώς γίνεται διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηροί κανόνες για να ανοίξουν νέοι τομείς εγκλήματος. Χρειάζεται ένταλμα μάλιστα για να αποφασιστεί ποια δεδομένα μπορούμε να χρησιμοποιηθούν και ποιοι είναι οι στόχοι για τις διάφορες αρχές. Όπως σας είπα, υπάρχει και η εποπτεία από τις εθνικές αρχές. Αυτές οι βάσεις δεδομένων τις ε, καλούμαστε να τις διαχειριστούμε. Και εδώ είναι μεγάλη η επένδυση. Άλλαξε ο κανονισμός το 2017 με μια ε, σε ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης των ε, δεδομένων. Παλιότερα είμαστε, βασιζόμασταν σε σύστημα, είμαστε, είχαμε, λειτουργούσαμε βάσει συστήματος. Τώρα λειτουργούμε βάσει στόχου. Κοιτάμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνει η Europol με τα δεδομένα που μοιραζόμαστε με διάφορες υπηρεσίες. Μπορούμε να τα μοιραστούμε, να τα χρειαστούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για ανάλυση, για θεματική ανάλυση, για λειτουργική ανάλυση και να τα χρησιμοποιήσουμε για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη. Αν τα κράτη-μέλη παραμένουν όμως ε, ιδιοκτησία της Εθνικής Αρχής και πραγματικά εμείς ε, συμμορφούμαστε και ε, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με τον τρόπο που επιθυμούν. Είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές. Για το ΣΥΣ τώρα. Ο νέος κανονισμός ετέθησε εφαρμογή το 2018 και πραγματικά μπορούμε να τα πάμε καλύτερα εδώ, όντως. Η εφαρμογή σε επίπεδο Europol θα είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη του 2019 και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθηθεί και ο δικός χάρτης για το IT. Η πρόταση για την διατήρηση των δεδομένων μέσω των εθνικών αρχών. Θα υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για το 5G. Δημοσιεύσαμε μία μελέτη για τις νέες τεχνολογίες. Και αυτά θα αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά οι αρχές επιβολής του νόμου. Ήταν σημαντικό λοιπόν να προετοιμαστούμε. Δημιουργήσαμε μια ομάδα εμπειροχνομόνων για θέματα επέκτασης των νέων τεχνολογιών. Επίσης, συνεργαστήκαμε και με, τις, ε, με τον οικονομικό κλάδο, τον μηχανικό κλάδο. Κάναμε μια πλήρη ανάλυση για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι μελλοντικέ απειλές από το 5G. Ένα από τα βασικά λοιπόν ζητήματα είναι ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να να ελέγχουμε την διακίνηση των δεδομένων. Προσπαθούμε λοιπόν και με τους συμπρεκνόμονες και στην Κυροπόλη να βρούμε μια λύση. Επίσης μιλώντας για νέες καινοτομίε που θα έχουν αντικτύπο στην εσωτερική ασφάλεια ή άμα κοινότητα της επαρμογής του νόμου θα πρέπει να συμμετέχει πιο πολύ για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας που θα προκύψουν από τις νέες τεχνολογίες αυτές. Αυτό το υποστηρίζουν όλα τα κρατημέλη και βλέπουμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα. Τι κάνουμε τώρα για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Europol. Αναπτύσσουμε μια πλατφόρμα κρυπτογράφηση στην Ίσπρα, στην Ιταλία, μαζί με το Κέντρο ε, Ψηφιακής Έρευνας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε πραγματικά κράβαδα, ότι αυτό είναι το μέλλον της ε, κοινότητας εφαρμογής του νόμου. Έχουμε επίσης γνώση του τι συμβαίνει στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα. Έχουμε επίσης και τους ακαδημαϊκούς ε, που προσπαθούν να βρουν ε, έξυπνες λύσεις προκειμένου να ε, μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες για τη Γαλλία, υπάρχει μεγάλη συνεργασία με τον δυτικό κλάδο, με τις τράπεζες, με τον αστυνομικό κλάδο με το δικαστικό κλάδο για να συζητήσουμε τα μεγάλα ζητήματα που ανακύπτουν σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις τράπεζες. Προσπαθούμε να δούμε πού έχει κενά το σύστημα, πού χάσκει, για να βρούμε κοινέ λύσεις. Σκοπός της ομάδας εργασίας για το Κέντρο Οικονομικού και Ψηφιακού Εγκλήματος ακριβώς αυτός είναι να βρει τις μελλοντικέ απαντήσεις και λύσεις προσπαθώντας να είμαστε πιο ενεργοί στα προβλήματα του μέλλοντος. Και φυσικά αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε πιο στενή συνεργασία με τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τις ε, ασυνόδευτους ανελίκους. Μεγάλο θέμα αυτό για μας και δεν ε, έχουμε αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη και δεν έχουν μπει αυτά σε μία μόνο βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά τους ε, ασυνόδευτου ανηλίκου. Εμεί, από πλευρά τη ε, Europol έχουμε μια υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση ανθρώπων. Εκεί κοιτάμε και το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων και πραγματικά θέλουμε στις επιχειρήσεις μας να το θέσουμε αυτό ως σημείο εστίασης στις επαφές με τα κράτη-μέλη. Όπως σας είπα, πάντα αναζητούμε νέες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα το οποίο κρύβεται πίσω από την παράνομη μετανάστευση και γι' αυτό ένα από τα βασικά στοιχεία είναι να υπάρχει ο αξιωματικός σύνδεσμο από τα κρατημέλη μαζί μας κάθε μέρα προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση διαρκώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, κυρία Ντεμπόλ και την ομάδα της Ευρωπόλ που βρίσκεται εδώ στο πάνελ, όχι μόνο για την λεπτομερέστατη παρουσίασή της, αλλά και για το ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και κατάφερε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που της έγιναν από τα μέλη της Επιτροπής μας. Θέλουμε να παραμείνει στενή η συνεργασία μας, γι' αυτό λοιπόν ε, θα σας ξαναδούμε και θα σας βλέπουμε συχνά. Να σας φίξω λοιπόν το χέρι και να σας αποχαιρετήσουμε διότι έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη που πρέπει να εξετάσουμε. Παρακαλώ καθίστε διότι έχουμε ένα τελευταίο θέμα το οποίο θα προσπαθήσω να εξετάσουμε σύντομα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί και Σήμερα λοιπόν έχουμε να εξετάσουμε και ένα επιπλέον σημείο που έχει να κάνει με την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη τη αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τι άδειε κυκλοφορία οχημάτων στην Ιρλανδία. Έχουμε να κάνουμε με εξέταση του σχεδίου έκθεση. οπότε σα παρακαλώ να καθίσετε για λίγο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Καθίστε γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ. Αφορά λοιπόν την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων για τις άδειες οχημά... κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία. Με την απόφαση αυτή το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δώσει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν δεδομένα με την Ιρλανδία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος. Αυτή η ανταλλαγή στοιχείων είναι βασισμένη στην απόφαση της συνθήκης του Προύμ έχει σταλεί μια επιστολή στο Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2019, όπου μας ζητείτε να γνωμοδοτήσουμε το συντομότερο δυνατόν, όχι μετά από τρεις μήνες, σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτία όμω των ευρωεκλογών η ημερομηνία αυτή έπρεπε να αλλάξει και να αναβληθεί. Τώρα λοιπόν η νέα ημερομηνία είναι 20 Σεπτεμβρίου 2019, αυτό το μήνα δηλαδή. Οι συντονιστέ συμφώνησαν να εξετάσουν την απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία του εσωτερικού μα κανονισμού Ακριβώ επειδή το ζήτημα αυτό επήγει και πρέπει να συμμορφωθούμε με τι υποχρεώσει μα. Μα έχει ζητηθεί λοιπόν η γνωμοδότηση από το Συμβούλιο και εγώ προσωπικά ήμουν εισηγητή. Πρότεινα λοιπόν να συμφωνήσουμε με την απόφαση του Συμβουλίου χωρί τροπολογίε. διότι είναι μια απόφαση η οποία θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και τη τρομοκρατίας. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορείτε να συμφωνήσετε. Υπάρχει, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Εσείς παρακαλώ. Ναι, εμείς θα θέλαμε να καταγραφεί και να γραφτεί στα πρακτικά η ένστασή μας, η διαφωνία μας με αυτό. Διαφωνείτε δηλαδή, ναι. Διαφωνούμε διότι συλλέγονται και ανταλλάσσονται δεδομένα με τρόπο δυσανάλογο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ωραία λοιπόν, καταλαβαίνω πως θέλετε να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά εκ μέρους της ομάδας της ΓΚΟΕ. Υπάρχει κάποια άλλη αντίρρηση. Όχι, νομίζω πως ε, θα έχουμε πλειοψηφία υπέρ της πρότασής μου. Και η ένστασή σας έχει μόνο διαδικαστικό χαρακτήρα. Αν το 10% των μελών το στηρίξουν, τότε θα αλλάξει αυτό. Αλλά δεν νομίζω να στηρίζει κανεί άλλο από εσά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το γνωρίζω αυτό, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να το πω. Ωραία, λοιπόν. Τότε μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο έκθεση. Ε, κύριε Σαρσαλέχο, θέλετε να πείτε κάτι, Όχι. Επομένως, η έκθεση εγκρίνεται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έγινε αυτό εγκαίρος για να προλάβουμε να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα που μας έχει δώσει το Συμβούλιο. Να σας κρατήσω μόνο για ένα λεπτό. Μου λένε ότι μας αφορά όλους το θέμα αυτό. Πρέπει να διαβάσουμε την ανακοίνωση σχετικά με τους εισηγητές που έχουν οριστεί σύμφωνα με την απόφαση των συντονιστών. Θα το διαβάσω πολύ γρήγορα λοιπόν. Ναι. Δεν το έκανα γιατί, είχε γιατί θα ακολουθούσε η φιλανδική παρουσίαση, αλλά θα το κάνω τώρα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό ακόμα. Εγώ, ο πρόεδρος, έχω οριστεί εισηγητή για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για τη Eurojust, για τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας. Επίσης, θα καταρτιστεί ψήφισμα για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Ο Πάουλο Ραντζέλ θα είναι εισηγητή για το σύστημα VIS. Η κυρία Γιατενμάκη για την ε, διαδικτυακή τρομοκρατία και σχετικό περιεχόμενο. Τέρον για έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα. Ο Γιάν Κρίστοφ για την έκθεση με τη στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση. Τάνια Φαγιόν τρίτες χώρες, οι υπήκοοι των οποίων εξαιρούνται από υποχρέωση θεώρησης, Κόσοβο δηλαδή. Χέρμαν Ίσελ για την πρόσβαση στα, του κοινού στα έγγραφα. Χέρμαν για την έκθεση στην ανταλλαγή πληροφοριών για κατάρτιση προσωπικού. Τάνια Φαγιών εσωτερική διαχείριση συνόρων και σχετικό ταμείο. Θεωρήσεις 2021-2027. Μόνικα Χολμάιερ, Εσωτερικό Ταμείο Ασφάλειας. Κατερίνα Μπαρλάι. Για τον κανονισμό Δουβλίνο, Κλοντ Μοραές. Οργανισμός ΕΑΣΟ. Λάουρα Φεράρα. Διεθνής προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοφίντφελντ, πρότυπα για την υποδοχή των διεθνούς προστασίας. Μπιόρκ, πλαίσιο επανεγκατάστασης. Ζίπελ, κανονισμός για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Κλοντ Μωραές. Η evidence. Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικέ διαδικασίε. Πίργκιτ Ζίπελ παρομοίω. Κλοντ Μωράες, μπλε κάρτα, Μετσόλα, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Λιχτενστάιν. για καταπολέμηση διασυνοριακού εγκλήματος και τρομοκρατίας. Ρομπέρτα Μετσόλα, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τους ίδιους σκοπούς. Σοφίντ Φέλντ, Συμφωνία Καναδά Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα PNR. Ρομπέρτα Μετσόλα. Διακανονισμός με την Ισλανδία για τη συμμετοχή της στην ΕΑΣΟ. Σίλβια Σπούρεκ. Προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την καταπολέμηση τη βία και της ένδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Ραντζέλ, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Βραζιλία για τι ε, θεωρήσει βραχία διαμονή. Βολάφ. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας για δράσεις της Frontex. Η ίδια συνάδελφος για την απόφαση του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαυροβουνίου. Επίσης για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στρίκ. Κοινά πρότυπα για την επιστροφή παρανόμως διαμένοντων από τρίτες χώρες. Ντέλμπος, κράτος δικαίου στην Ουγγαρία και τέλος Ντέλη για τον κανονισμό ενός κανονισμού που έχετε μπροστά σας, δεν διαβάζω τώρα τον αριθμό του, για την ε, παραποίηση. Συμφωνείτε με αυτούς ε, τους εισηγητές και τις εισηγήτριες. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν για σήμερα και να σας ενημερώσω ότι θα συνεχίσουμε με κοινή συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 12.30 λέει ο πρόεδρος. Στις 2.30 στην αίθουσα ASP1G3. Όμως, μέχρι τις 3.30 και για τις τρεις επόμενες ώρες συνεχίζουμε εδώ. Όχι στον, στο δύο όροφους κάτω, στον πρώτο. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε αργότερα.